Καλή μέρα. Όλοι, είστε, όλοι όσοι είστε εδώ στην αίθουσα και όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του διαδικτύου. Θα συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας ε, που ξεκίνησε χτες. Θα ήθελα να καλωσορίζω τον ε, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, τον κύριο Αλέξης Γκόστελ θα μας ε, παρουσιάσει την ε, απόδοση του έργου και τις ε, επιτυχίες του κέντρου το 2018 και το προβλεπόμενο έργο του για το 2019. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Γκόστελ για μια σύντομη ή λιγότερο σύντομη παρουσίαση, εξαρτάται τι, από το τι θέλετε να μας πείτε. Και ενδεχομένως μετά θα πάρουμε ερωτήσεις από εσάς. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά μου έρχομαι στην Επιτροπή Λίμπερ να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες και το έργο του κέντρου το 2018. Όπως σας έλεγα και πριν ξεκινήσουμε, θα θυμάστε πως όταν ανέλαβα τα καθηκόντά μου ως διευθυντού του κέντρου, είχα ε, προτείνει προτείνει ε, ο προγραμματισμός να γίνει λίγο πιο νωρίς όχι, μέσω, όχι ανάμεσα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο που γίνεται κάθε φορά αλλά πιο νωρίς και χαίρομαι που η Επιτροπή σας μας στήριξε οπότε τώρα ο προγραμματισμός και η παρουσίαση γίνεται γύρω στις 15 Φεβρουαρίου το νωρίτερο που, γίνεται, που μπορεί να γίνει για να είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε ε, στοιχεία και για τα οικονομικά και δημοσιονομικά και το, για το πώς καταφέραμε να υλοποιήσουμε τις διάφορες προτεραιότητες του κέντρου. Όπως ε, λέει και το εξώφυλλο, είμαστε προσιλωμένοι στο έργο μας να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ε, αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και σε όλο τον κλάδο. 48 εκθέσεις ε, δημοσίευσαμε πέρσι. Υπογράψαμε ή συνυπογράψαμε 23 επιστημονικά 23 επιστημονικές εργασίες πιο πολύ δηλαδή από ότι το 2017. Ε, σαράντα 40 εκθέσεις αναχώρα είναι ο νέος τρόπος τον οποίο έχουμε επιλέξει για να παρουσιάζουμε τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην χρειάζεται τα κράτη-μέλη να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα. Εμείς τα παίρνουμε, παίρνουμε τις πληροφορίες των κρατών μελών, προσθέτουμε γραφικές παραστάσεις και συγκρίνουμε το, την κάθε χώρα με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά δύο ειδικέ δημοσιεύσει. Μία για πρώτη φορά για την ε, ιατρική χρήση προϊόντων της κάναβης. Σας είχαμε, είχαμε ενημερώσει από πέρσι. Πολύ σημαντικό γιατί είχε σχέση και με το, ε, ψήφισμα ε, του Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβουρού. Ε, συνεργαζόμαστε και με την ε, υπηρεσία φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν είμαστε ρυθμιστική αρχή, αλλά η ιατρική χρήση των προϊόντων της κάναβης βρίσκεται στην τομή της πολιτικής για, τη για τα ναρκωτικά και στον, του κλάδου της, ε, των φαρμάκων. Οπότε για πρώτη φορά δίνουμε ένα πανόραμα ε, των διαφόρων δημοσιεύσεων που έχουν γίνει, αξιολογήσεων κλπ. και δίνουμε πληροφορίες για το πώς μπορούμε να, να κατατάξουμε τα πορίσματα. Υπάρχουν κάποιες α, αρνητικές κάποια αρνητικά πορίσματα από έρευνες, οι οποίες όμως συνήθω βασίζονται σε πολύ μικρό αριθμό, ε, πολύ μικρό δείγμα, πολύ μικρό αριθμό ε, ατόμων που συμμετεχόντων, οπότε είναι δύσκολο ε, να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου τύπου έρευνες να ξέρουμε σε τι στοιχεία βασίζονται. Δεν είναι ότι είναι λαθασμένα τα αποτελέσματα απαραίτητα, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε περισσότερη διερεύνηση. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία υπογραμμίζει και το ίδιο το ψήφισμα, πόσο ξέρω. Δεύτερο πυλώνας της ε, υλοποίησης στρατηγικής μας είναι η αύξηση της παρουσίας μας, της ορατότητάς μας. Αυξήσαμε κατά 28% τον αριθμό των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή το 2018, καταγράφηκαν πάνω από 1.360.000 άτομα που επισκέφθηκαν τον ιστοχώρο μας και μιλάμε για μοναδικούς επισκέπτες. Έτσι δεν πρόκειται ο ίδιος, δεν πρόκειται για κάποιον ο οποίο επισκέπτεται διαφορετικές σελίδε. Επίσης, αυξήσαμε κατά 70% ε, τα downloads των διαφορών βίντεο που παράγουμε. Αυτό είναι κάτι καινούριο στην επικοινωνιακή μας στρατηγική. Ακολουθούμε τα πιο πρόσφατα trends που είναι λιγότερο κείμενο, ε, λιγότερη σύνδεσμοι και αύξηση του ακουστικού υλικού. Έχουμε για παράδειγμα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για το τι σημαίνει ε, ε, ε νομιμοποίηση. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Κάθε Ιούνιο σας υποβάλλουμε μία έκθεση. Ε, η έκθεση αυτή πέρσι ε, γινόταν download κάθε 10, μία φορά κάθε 10 λεπτά. Ως στρατηγική επίσης ε, έχουμε την διευκρίνηση και την ενίσχυση των υπηρεσιών προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους. Έχουμε συνεισφέρει σε, με τη γνώμη μας 60 διεθνείς ε, συναντήσεις. Σε πολλές φορές στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Προεδρία, για παράδειγμα στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων ή κατά την προετοιμασία της ε, ε, παρακολούθηση της UNCAST, δηλαδή της Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για το, τα ναρκωτικά κλπ. Έχουμε συμμετάσχει σε πάνω από 300 διαφορετικές, σε πάνω από 300, 300 εκδηλώσεις τεχνικής ε, και επιστημονικής φύσεως και τέλος έχουμε εξυπηρετήσει 45 πέντε αιτήματα από θερμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εξυπηρετούνται σε μια προθεσμία μικρότερη των δύο εβδομάδων. Για παράδειγμα, μας ρωτάνε Ιράν, τι γνωρίζουμε για την κατάσταση του, του θέματος των ναρκωτικών στο Ιράν ή για τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη χώρα. Επίση, εξυπηρετούμε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν έρχονται σε εμά με αιτήματα ή ερωτήσει. Και όλα αυτά έγκαιρα και γρήγορα. Μέσα στις προθεσμίες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες στην Ευρώπη. NPS. Ε, τα τελευταία 5-10 χρόνια έγινε μια έκρηξη, εκρηκτική αύξηση τέτοιων ουσιών ε, που εντοπίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκθετική αύξηση. Ε, η τάση βέβαια είναι μειωτική τα τελευταία χρόνια, λίγο μειωτική. Πέρσι εντοπίσαμε 55 νέες ουσίες, δηλαδή μια, μια εβδομάδα κατά όρο 392 συνολικά ουσίες έχουν ε, εντοπιστεί. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο νούμερα. 55 είναι ο αριθμός των ουσιών που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πέρσι. 392 είναι συνολικά οι ουσίες NPS που έχουμε εντοπίσει στην αγορά μέχρι, ε, ε, που εντοπίσαμε πέρσι ε, στην αγορά, 392, 55 ήταν οι καινούριε, πάνω από 750 είναι συνολικά οι ουσίε MPS που έχουμε εντοπίσει στα περασμένα χρόνια. Δηλαδή κάποιες εξαφανίζονται, μετά ξαναεμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται, οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι διαφορέ. 392 ουσίε εντοπίστηκαν συνολικά πέρσι, εκ των οποίων 55 ήταν καινούριε, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Επίση πέρσι ε, κάναμε δύο αξιολογήσεις κινδύνου και θέσαμε υπό, σε, ε, και το Συμβούλιο θέσε σε ε, παρακολούθηση τέσσερις νέες ουσίες με βάση αυτές τις μελέτες αξιολόγησης κινδύνου που έχουμε κάνει. Επίσης έχουμε τη νέα νομοθεσία για τις ουσίες NPS, η οποία ε, θα τεθεί σε εφαρμογή και σύμφωνα μάλιστα με τις απαιτήσει ολοκληρώσαμε την διαδικασία της ε, ε, επεξεργασίας των κανόνων συνεργασίας με τις ε, πέντε συναρμόδιες, με, τα πέντε, τις πέντε συναρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Τώρα, η επίδοση του, κέντρου μας. Όπως σας έχω πει, ε, θέλουμε να να ονόμαστε με τους κανόνες, να είμαστε αποτελεσματικοί, διαφανείς και έχουμε καθορίσει ένα σύνολο προτεραιοτήτων. Θέλουμε, ανάλογα με, τις, ε, με τους πόρους που διαθέτουμε, να τους ε, κατανέμουμε σύμφωνα με αυτές τις προτεραιότητές μας. Η απόδοση μας είναι εξαιρετική. Οι προτεραιότητες L1 είναι για αυτές τις οποίες θέλουμε να φτάσουμε στο 100%. Πέρσι Εφέτος, πέρσι το 18, δηλαδή ήμασταν στο 95%. Είχαμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την νέα βάση δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ψυχοδραστικέ ουσίε τι NPS. Ελπίζουμε ότι το τρέχον έτος θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες αυτές. Έχουμε το πρώτο κομμάτι της βάσης δεδομένων και ε, ήδη κάνουμε τους, τα πρώτα τεστ. Οι προτεραιότητες L2 αφορούσαν δραστηριότητες ε, στις οποίες είχαμε ένα στόχο 80%, έχουμε φτάσει 95% περισσότερο από πέρσι και για, το, για τις προτεραιότητες L3 είχαμε στόχο 50%. Οπότε αν πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές, αν οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, σίγουρα δεν θα κόψουμε κονδύλια από τις ε, προτεραιότητες Ελένα, αλλά από τις υπόλοιπες. Καλές οι επιδόσεις μας λοιπόν. Από τους 200 περίπου στόχους, μόνο δύο ακυρώθηκαν και για καλούς λόγους, διότι άλλαξε η πραγματικότητα. Τώρα, εξωτερική αξιολόγηση ήταν το βασικό, η βασική στιγμή κρίσης για μας πέρσι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Γιατί μπορούμε να σας πούμε ότι το Νοέμβριο, Δεκέμβριο πέρσι ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση και οι συνάδελφοι από την Κομισιόν θα το επιβεβαιώσουν. Νομίζω ότι είναι τα καλύτερα από αποτελέσματα που είχαμε ποτέ από εξωτερική αξιολόγηση. Και το εκτελεστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο, συγγνώμη, και εγώ είμαστε πολύ περήφανοι. Βλέπω ότι αναγνωρίζεται η τεράστια προσπάθεια που κάναμε κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ιτίας μου για να βελτιώσουμε την παρακολούθηση της απόδοσης και της εκτέλεσης, καθώς επίσης και την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής που μας επιτρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο ε, για ποιον εργαζόμαστε, ποια είναι η προσθέμενη αξία μας, τι περιμένει ο κόσμος από μας. Τεράστια προσπάθεια λοιπόν και θέλω δημοσίως να ευχαριστήσω τους αδέλφους της ε, Κομισιόν εκ μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου γιατί η δουλειά ήταν τεράστια. Για πρώτη φορά η αξιολόγηση δεν κάλυψε μόνο τους δείκτες απόδοσης αλλά και τον αντίκτυπο του έργου μας. οι δύο βοηθοί μου που βοήθησαν την Κομισιόν σε αυτήν την εξωτερική αξιολόγηση χρειάστηκαν να παράσχουν και να εξηγήσουν στην Κομισιόν 250, 250 με 280 φακέλους. Το σημαντικό επίσης είναι ότι ένα κομμάτι της αξιολόγησης αυτής αφιερώθηκε στο ποιε είναι οι ανάγκες διεύρυνσης των καθηκόντων του κέντρου. Έγιναν πολλές προτάσεις και τις συζητήσαμε το Δεκέμβριο με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν αλλά πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, γιατί πρόκειται για μια σημαντική μετάβαση. Η δική σας επιτροπή προφανώς θα παίξει σημαντικό ρόλο και εγώ πολύ ευχαριστώ να ξαναέρθω όποτε το επιθυμείτε για να απαντήσω σε ερωτήσεις για το πώς μπορεί να αυξηθεί η ορατότητά μας, πώς μπορεί να τροποποιηθεί η εντόλη που μας έχει δοθεί. Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για συμμόρφωση, μιλάμε για απόδοση, αλλά είναι πολύ σημαντική και η οικονομία, τα οικονομικά στοιχεία. Για τρίτη σε σειρά χρονιά καταφέραμε να φτάσουμε σχεδόν στο 100% της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Είναι μοναδικό αυτό στην ιστορία μας, 99,98%. Αυτό που αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πλέον ευελιξία στον προπολογισμό μας. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τις, την εκτέλεση των πληρωμών. Από το 94,5% φτάσαμε στο 98,02% φέτος. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα βέβαια αλλά είναι αδύνατο να φτάσουμε το 100% γιατί δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τους μισθούς. Οπότε ε, αυτά τα δύο νούμερα είναι, ε, ταιριάζουν μεταξύ τους. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων C8, που δεσμεύονται ένα χρόνο, αλλά οι τελικές πληρώμεις γίνονται τον επόμενο χρόνο, βρισκόμαστε στο 94,2%. Ε, δεν είμαστε το 100% γιατί μερικές φορές τα κράτη-μέλη δεν δίνουν στα σημεία επαφή μας τα ποσά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Οπότε ε, τα ποσά τα οποία δεν αναλώνονται εδώ ε, μεταφέρονται αλλού δεν χάνονται ε, και μόνο 25-30 χιλιάδες ευρώ θα επιστρέψουν στον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πάντως η απόδοση αυτή είναι πολύ καλή. Η Επιτροπή σα και η Κομισιόν παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση, το γνωρίζω. Και εμείς οι ίδιοι παρακολουθούμε την εφαρμογή των συστάσεων του Ελεκτικού συνεδρίου και της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου και πέρσι πέραν της εξωτερικής αξιολόγησης έγινε και μια, ε, ένας ε, εσωτερικός έλεγχος για τις ε, διαδικασίες δημοσίευσης του κέντρου μας και μπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. αυτό είναι το, ο καρπός προσπαθειών τριών ετών. Όταν ανέλαβα, η η ε, κατάσταση των σχέσεων με το, ε, με το ελεκτικό συνέδριο ήταν κρίσιμη και νομίζω ότι ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη. Αφιερώσαμε χρόνο και εξομαλύναμε τις σχέσεις μας. Η υλοποίηση ορισμένων συστάσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, επιχειρηματική αρχιτεκτονική, ε, μας βοήθησαν πολύ. Θα επανέλθω αν έχουμε χρόνο. Τι, έγινε, τι καινούριο έγινε πέρσι και θα συνεχιστεί και φέτος, είναι ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μας και των μας, δημοσιεύσεών μας ε, αφιερώθηκαν στο να ενημερώσουμε τους πάντες για το τι συμβαίνει με την κάναβη, τι το πίμαχο υπάρχει, ποιε είναι οι προκλήσει για το μέλλον. Συνεπώ ε, ε, ετοιμάσαμε μια δημοσίευση με ερωτήσεις και απαντήσεις. Στις 5 Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε, δημοσιεύσαμε ε, μια μελέτη για την ιατρική χρήση της κάναβης και των ε, παραγόντων της, των υποπροϊόντων της, και ήδη είχα εξηγήσει από πέρσι ότι δεν θεωρούμε πως η όρος ιατρική χρήση είναι ο πιο καλός, γιατί στην ιατρική ε, δεν μιλάμε για φυτά, μιλάμε για συγκεκριμένες ουσίες και αυτές οι ουσίες είναι που έχουν ιατρική χρήση, όχι το ίδιο το φυτό ή το ζώο. Οπότε θα πρέπει να μιλάμε για ιατρική χρήση των ουσιών που περιέχονται στην κάναβη, των καναβινοειδών. Επίσης, ε, οι δημοσίευσεις μας για, τις, ε, για τα νέα, για τα πιο επίγοντα νέα, ε, πηγαίνουν πλέον σε διπλάσιους συνδρομητές. Ε, δεν δίνουμε βέβαια εκεί ζεστές ειδήσει, επικέρες ειδήσει. Πρώτα εξετάζουμε την κατάσταση, δεν πρόκειται να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε φήμη ακούγεται, τρελή φήμη ακούγεται. Ε, εξετάζουμε, μελετάμε και μετά δημοσιεύουμε τα πορίσματά μας μέσω αυτής της δημοσίευσης. Βγάζουμε συμπεράσματα, ενημερωνόμαστε και μετά ενημερώνουμε και εμείς το κοινό μας. Και έχουμε και δύο καινούρια προϊόντα για φέτος. Πρώτον, μια δημοσίευση ε, για προϊόντα της κάναβης ε, χαμηλά σε THC, καναβιόλι, THC, Μας ζητήθηκε να διευκρινίσουμε τι είναι αυτά ακριβώς τα προϊόντα και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερη δημοσίευση, ίσως μια διπλή δημοσίευση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αλλαγών στις πολιτικές για την κάναβη. Ε, λαμβάνοντας υπόψη τις, ε, τα αριθμιστικά μοντέλα της αγοράς, γιατί εκεί μερικές φορές επικρατεί σύγχυση. Αν δείτε την πολιτική των διαφορετικών πολιτιών, των ΗΠΑ, της Ουγγάης και του Καναδά, καμία από αυτές δεν έχει νομιμοποιήσει την κάναβη με τον ίδιο τρόπο. Ε, δεν θα βρείτε δύο χώρες που να έχουν πάρει τα ίδια μέτρα. Οπότε υπάρχουν επιλογές οι οποίες πρέπει να γίνουν ε, και ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για τις επιλογές αυτές. Έχουμε για το 2019 δύο εκδηλώσεις και δημοσιεύματα. Έχουμε την τρίτη έκδοση, της, ε, την τρίτη διάσκεψη ε, της διάσκεψη, ε, τρίτη διάσκεψη της Λισαβόνας. Είναι η πιο σημαντική διάσκεψη στην Ευρώπη για τα ναρκωτικά. Πάνω από 1.300 συμμετέχοντες ε, έλαβαν μέρος από πάνω από 60 χώρες την δεύτερη διάσκεψη που έγινε. Στη φετινή τρίτη διάσκεψη θα έχουμε μία συνεδρία θα είναι αφιερωμένη στο μέλλον. Θα προσπαθήσουμε, όπως είχε αποσχεθεί πριν από 1,5 χρόνο, να δούμε ποιες θα είναι να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από πλευρά πολιτική, δηλαδή πρόληψη, καταστολή κλπ. για το μέλλον. Και μετά, και νομίζω ότι εδώ τελειώνουμε, όπως κάνουμε τα τελευταία τρία χρόνια τον, και το κάναμε και το πέρσι, ε, θα δημοσιεύσουμε μαζί με την Ευρωπόλ το Νοέμβρη ε, την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Αγορά Ναρκωτικών. Θέλω να ε, ευχαριστήσω το συνάδελφο διευθυντή της Europol που μας βοηθάει και συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με όλη αυτή τη συνεργασία ίσως θα έπρεπε να ε, συστεγαζόμαστε κιόλας να σα πω την αλήθεια γιατί πραγματικά έχει, υπάρχει πολλή μετακίνηση πληροφορίε από τη μία στην άλλη. Ε, η, Ευρω... η Ευρωπόλ επίσης πέρσι ε, ε, αποφάσισε να δίνει περισσότερο βάρος στο θέμα των ναρκωτικών από το 2000. 16 υπολογίζεται ότι η αγορά ήταν 28-30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν ερχόταν σε αυτό το ποσό, κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάμε για ποσά τα οποία τροφοδοτούν πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Δεν αφορά δηλαδή μόνο ναρκωτικά, ε, αυτά τα ποσά πηγαίνουν και αλλού τελικά, σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως αυτή είναι μία από τις τελευταίες συναντήσεις με αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους όλου του προσωπικού του κέντρου, του προκατόχου μου και μου του ιδίου. Α, ε, ε, ε ξεχάσα αυτό το, αυτή τη διαφάνεια ε, και δεν θα μου το συγχωρέσουν συνάδελφοι μου. Ε, να τελειώσουμε τι ευχαριστίες καταρχήν προς την Επιτροπή σα. Η στήριξή σας ήταν κρίσιμη για μας όλους και για μένα. Όταν είχε γίνει η ακρόαση μου, η, Επιτροπή μου είχε ζητήσει να βελτιώσω την απόδοση ε, ε, του κέντρου μας και μετά να ζητήσω λεφτά. Μετά από τρία χρόνια βελτίωσης ε, της απόδοσης μπορώ να πλέον να μιλήσω και για χρήματα. Οπότε ένα από τα προβλήματα που έχουμε ως παλαιά υπηρεσία προς παλαιό, ως παλαιό κέντρο. Έχουμε κλείσει 25 χρόνια. Ε, ο κανονισμός που μας αφορά υιοθετήθηκε πριν από 26 χρόνια. Έχει σχέση με τον τίτλο 1 του προπολογισμού ε, που είναι το μισθολογικό κόστος που φτάνει στο 70% του προπολογισμού μας. Κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη αύξηση χωρίς καμία απόφαση από μένα ή από το Διοικητικό Συμβουλίο, οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη αύξηση ε, αναπροσαρμογή των μισθών επηρεάζει πάρα πολύ τις δραστηριότητε μας. Ήδη είχαμε προβλήματα με την αύξηση του ενοικίου μας. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ και 25 η Νοεμβρίου πέρσι χρειάστηκε να κόψω 1,3 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να παραμείνω μέσα στα όρια του προπολογισμού μας. Το 1 εκατομμύριο οφειλόταν στους, στην αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των μισθών και του ενοικίου μας. Το κρίσιμο έτος θα, ήταν το 2020. θα είναι το 2020. Γιατί, Γιατί οι υπηρεσίε τη Κομισιόν μας αναφέρουν ότι πιθανότατα θα γίνει μία ακόμα αύξηση των μισθών. Έστω και ήπια να είναι, μαζί με την διόρθωση που γίνεται, με βάση το βιωτικό επίπεδο, στην Πορτογαλία ο βασικός μισθός αντιπροσωπεύει το 77-78% του ίδιου προσωπικού που θα δούλευε αν δούλευε στις Βρυξέλλες. Ε, και με την αλλαγή του συντελεστή εξαιτία τη μεταβολή του βιωτικού επίπεδου στην, ε, στην Πορτογαλία, ε, θα έπρεπε να, ξανα, να βρούμε άλλο ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω πού θα τα βρω. Δεν ξέρω πού θα μπορούσαμε να τα βρούμε. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την καλύτερη εξωτερική αξιολόγηση που είχαμε ποτέ. Δηλαδή κάθε ένα ευρώ, κάθε ένα λεπτό του ευρώ δαπανάται σωστά και επιπλέον, πιθανότατα θα μας δοθούν και περισσότερες αρμοδιότητες, διότι έχουμε και καινούριου κινδύνους. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανεβάσουμε τον πύχη. Δεν θα έλεγα ότι θα υποχρεωθούμε να κλείσουμε, αλλά θα, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε μία ακόμα περικοπή με αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε επιπλέον περικοπές. Και νομίζω ότι τα ε, οικονομικά μας στοιχεία το στηρίζουν αυτό που λέω. Η καλή είδηση είναι ότι με τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσαμε να υποβάλουμε ένα αίτημα για μεγαλύτερα ποσά από αυτά που προβλέπονται στην διαπραγματευσή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης η άλλη καλή είδηση είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Home μας στηρίζει στεναρά που ήδη αξιολόγησαν ε, το αίτημά μας, θεωρούν ότι πράγματι πρόκειται για ε, αύξηση που θα αφορά την επιβίωση του κέντρου μας, όχι για την αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Εμείς δεν ελέγχουμε το μισθολογικό κόστος, ούτε το ενίκιο. Γιατί οι μισθοί έρχονται στο, αν, έρχονται στο 70% του προπολογισμού μας. Η εξωτερική αξιολόγηση ανακάλυψε ότι έχουμε έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην υπηρεσία, στο κέντρο μας, για την ανάλυση της κατάστασης. Οπότε τα προηγούμενα χρόνια με την υποστήριξη της Επιτροπής Λίμπε και της Κομισιόν ε, ο προπολογισμό αυξήθηκε, έχει αυξηθεί και έχει αυξηθεί και το προσωπικό. Ε, Βέβαια, ε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν μόνο 100 άτομα στην Ευρώπη που έχουν αυτές τις ικανότητες, οπότε εμείς τους χρειαζόμαστε. Οπότε δεν ζητάμε μεγαλύτερο, περισσότερο προσωπικό, ζητάμε απλώς να μας επιτραπεί να δουλέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μπορείτε να βοηθήσετε Εσεί προετοιμάζετε ασφαλώ, προετοιμάζεστε για τι επόμενε εκλογέ ή προσχέσετε σε προεκλογική εκστρατεία. Καλή επιτυχία. Και ελπίζουμε θα συνεργαστούμε και με την καινούρια σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμω συζητώνται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, το πολυμετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν νέε ανάγκε για έρευνα ε, σε θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά. Είναι ένα από τα θέματα του ψηφίσματος για την κάναβη. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά μην φανταστείτε ότι τελειώνει εδώ η δουλειά σα. διότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σα και φέτο. όπως μπορέσετε. Να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει τουλάχιστον να λειτουργούμε όπως σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς ευρωβουλευτής τον λόγο, αλλά εγώ ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Ε, να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ αναλυτική η παρουσίασή σας ε, και μας θυμήσατε διάφορες πτυχές των εργασιών σας, ε, τις ε, εκθέσεις ε, που εκπονείτε, τα αιτήματα που λαμβάνετε, η προσέγγιση των πολιτών, η ευαισθητοποίηση. Η εντύπωση λοιπόν που μας δώσατε είναι ότι είναι πολύ χρήσιμος ο οργανισμός και ότι τα χρήματα που δαπανώνται για τον οργανισμό αυτόν είναι απαραίτητα και δαπανώνται με σωστό τρόπο. Στο τέλος αναφερθήκατε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας σε μια κοινή πρόκληση, διότι θα αυξηθούν οι δαπάνες όχι μόνο για το δικό σας οργανισμό. Γενικά απαιτώνται περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει η απαραίτητη χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν συζήτηση σχετικά με την νέα χρηματοδότηση από πλευρά των κρατών μελών ε, ή για νέους ίδιους πόρους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση γενικά, αλλά και για τον οργανισμό σας που κάνει πολύ καλή δουλειά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις μελλοντικέ εργασίες ε, του οργανισμού σας και καλή επιτυχία και σε εμά στις επικείμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ και πάλι σήμερα για την παρουσίασή σας και κάθε επιτυχία στις μελλοντικέ σας εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε μια μελέτη για την κάναβη και την νομοθεσία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και η συζήτηση για την κάναβη θα συνεχιστεί στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, περνάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. που είναι η κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Θα ακούσουμε τον συνάδελφο Μάμικινς, που είναι η συγητής ε, και έχει να κάνει το θέμα με υποβολή αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με τι διαπραγματεύσει. Κύριε Μάμικιν, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω γνωρίζετε, έχουμε τον κανονισμό για την κυκλοφορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Μετά από δύο τριμερείς διαλόγους και δύο τεχνικές συζητήσεις τους τελευταίους μήνες καταλήξαμε σε συμφωνία. Το κείμενο εγκρίθηκε στην Κορεπέρ την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και τις ομάδες τους, ε, την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ για την καλή συνεργασία. Και όσον αφορά την ουσία του ενοποιημένου κειμένου, έχει πολύ ισχυρότερο ρυθμιστικό αντίκτυπο σε σχέση με τον κανονισμό του 2013. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και την ε, σωστή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ξεκαθαρίσαμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τους διάφορους ορισμούς. Ε, έχουμε πιο ισχυρές διατάξεις για τον εντοπισμό ε, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών αγορών. Ε, επίσης, ευαισθητοποίηση του κοινού για ε, τις πολύ επικίνδυνες ουσίες όπως είναι το οξύ. ενώ στην Ουγγαρία και στην Γερμανία έχουν καταργηθεί οι παλιές ρυθμίσεις για τα εκρηκτικά. Επίσης ε, προβλέπεται μια διαδικασία ε, ε, ενημέρωσης του επόμενου κρίκου στην αλυσίδα εμπορίου. Και επίσης Έχουμε τώρα ένα τελικό κείμενο το οποίο λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες όσον αφορά την ασφάλεια και τους στόχους της ενιαίας αγοράς ο οικονομικός αντίκτυπος του κανονισμού αυτού στην χημική βιομηχανία και άλλους οικονομικούς φορείς είναι αμεληταία σε σχέση με τα ωφέλη ως προς την ασφάλεια. Φυσικά στις διεθνείς διαπραγματεύσει έχουμε καταλήξει σε ισορροπημένο κείμενο, ωστόσο θα ήθελα το Συμβούλιο να δώσει περισσότερη προτεραιότητα ε, στις επιχειρήσεις ε, από ότι στην ασφάλεια σε κάποιους ε, τομεί, όπως για παράδειγμα τον περιορισμό της κυκλοφορίας στην αγορά των κάποιων εκρηκτικών υλών. Επίσης, σε περίπτωση νέων στοιχείων μπορούν να ληφθούν νέα μέτρα από τα κράτη-μέλη. Αυτό συνεχίζει να ισχύει και με τον νέο κανονισμό, παρότι ο στόχος του είναι να ε, πετύχουμε περισσότερη εναρμόνιση. Αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού θα γίνει πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή. Ελπίζω όμως το Κοινοβούλιο να μπορεί στο μεταξύ να λάβει κάποια προκαταρτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Είχαμε επιθέσεις στις Βρυξέλλες και το Μάνσεστερ το 2016 και 2017 και αλλού και γι' αυτό το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να παρουσιάσει αποτελέσματα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Ασφαλείας. Επιμένουμε στις προτεραιότητές μας για εναρμονισμένους ε, κανόνες ε, και για αντίδραση στην τρομοκρατική απειλή, ε, αλλά και διασφάλιση των συμφερόντων των οικονομικών φορέων. Πιστεύουμε ότι η λίστα πρέπει να είναι αναλογική σε σχέση με τις απειλές ως προς την ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε και ο κανονισμοί όπως ο παρόν αποτελούν ε, ε, απαραίτητο εργαλείο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συνεργασία σας, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ε, και κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έκθεση. Ορισμένοι σκιώδεις είναι εδώ. Ο κύριος Ντεχόφσκι νομίζω θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες. Σε ό,τι αφορά την περιγραφή της κατάστασης, δεν με ικανοποίησε αυτό που είπατε για πολλά. Η συμφωνία είναι πολύ καλή, πολύ καλή, ε, τριμερί, καλές τριμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τις ομάδες τους για μια εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του τι χρειάζεται από την πλευρά των πληροφοριών από οικονομικούς παράγοντες και του έργου των αστυνομικών αρχών αφετέρου αλλά και των υπεύθυνων ασφαλείας. Εγώ νομίζω ότι βελτιώνουμε την ασφάλεια και λαμβάνουμε παρκώς υπόψη τις ανάγκες των οικονομικών φορέων. Άρα είναι σαστή, σωστή ισορροπία σε ό,τι αφορά την έκθεση των προδρομών, τη αγορά σε προδρομής ουσίας εκρηκτικών υλών. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία. Νομίζω ότι συνολικά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Θέλω λοιπόν να υποστηρίξω αυτή τη συμφωνία. Παραλαμβάνω είναι πολύ ισορροπημένη πρόταση και θα δώσει λύσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα δίστανται οι πολιτικέ απόψει μετά το αποτέλεσμα κάποιου μέρου διαλόγου, όπω συνήθω. Η Ναταλή ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ω πρόεδρος ε, της Ειδική Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ως σκιώδης εισηγητρία για τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα, σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Μάμικιν, για το ποιοτικό έργο, γιατί την βικονούς και διαπραγματεύτηκε με πολύ ταλέντο πυκνότητα και ομαλή ροή της ε, διαπραγματεύσεις πάνω σε ένα τεχνικό απριόρι θέμα. Και τον ευχαριστώ γιατί βοήθησε σε πολύ καλό ρυθμό να προχωρήσει ο φάκελος και να περατωθούν οι εργασίες ε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα πριν το τέλος της θητείας. Ήταν σημαντικό και δύσκολο να βρεθεί μια χρυσή τομή, ιδίω με την πλευρά της βιομηχανίας, αλλά νομίζω ότι το πετύχαμε. Και νομίζω ότι περισσότεροι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν με το τελικό κείμενο. Είναι σαφές αποτελεσματικό το κείμενο και σε ό,τι αφορά το καρθόδε ζήτημα, τη συμπέριληψη δηλαδή των ε, γραμμικών ε, πωλήσεων, ε, είναι ένα θέμα που μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα ιδίως στη δική μου ομάδα σε ό,τι αφορά την διάδοση των πληροφοριών. Νομίζω ότι και εκεί καλά τα καταφέραμε και θα παροτρύνω, δεν ξέρω εσείς ε, τι είπατε ακριβώ, ε, κύριε Μαμίκινς, είπατε να μην είναι μοναχικά βαράρδες τα κράτη-μέλη. Το συντομότερο δυνατό λοιπόν πρέπει να υπάρξει έναρξη ισχύω για τον κανονισμό που θα καταφέρει να ανακόψει την απειλή αυτή της τρομοκρατίας. Ως Γαλλίδα ε, ιδιαίτερα τονίζω το θέμα της ε, τεχνολογίας και που και αυτή από τους τρομοκράτες στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους και συζητητές και συμφωνώ ακόμα και στον τομέα των εκρηκτικών υλών. Βλέπουμε να εμφανίζονται νέες ύλε και θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι χρησιμοποιούνται και σε νόμιμους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν πάντα να γνωρίζουμε ποιοι, ποιες ύλες είναι απαραίτητες για τις διάφορες χρήσεις και να τις ελέγχουμε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η νέα νομοθετική πρόταση θα οδηγήσει σε περισσότερη σαφήνεια και περισσότερο έλεγχο στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους κοιόδες εισηγητές για τη δουλειά τους και που ε, έκαναν δυνατή, την κατέστησαν δυνατή τη λήψη απόφασης πριν την επόμενη θητεία. Ε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ψηφοφορίες ε, σήμερα το πρωί. Θα ψηφίσουμε στις 11 και 4 το θέμα αυτό και ε, πιθανότατα να πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Συνάδελφοι, θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής μας που θα περάσει στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, διάλειμμα ο λίγων λεπτών. Δύο λεπτά διάλειμμα και ευχαριστώ θερμά και την κυρία Σίπελ που προείδρευσε το πρωί. Σας ευχαριστώ. Okay, Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την ε, υπομονή σας. Περιμέναμε λίγο γιατί μας είχαν πει δύο-τρει συνάδελφοι ότι θα έρχονταν ειδικά για το σημείο αυτό της μερισιάς διάταξης ε, για να ακούσουν τον Υπουργό. Θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου την κυρία Ζίπελ η οποία με αντικατέστησε όσο είχα αυτή τη συνάντηση με το Σύμβολο για την Ουγγαρία την ευχαριστώ, Μπίρκιτ, σε ευχαριστώ και για χθε και για σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μα τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική τη Ελλάδο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που μας αφιερώνει χρόνο η Επιτροπή μας φυσικά παρακολουθεί του σύνεγγυς και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κατάσταση στην Ελλάδα μέσω κάποιων επιτόπιων αποστολών, ανταλλαγών απόψεων που αφορούν θέματα χρηματοδότησης. Επίσης λαμβάνουμε τακτικά ενημέρωση για την κατάσταση στα hot spot και την υλοποίηση της ε, ε, συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μετά την τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε τον Ιούνιο, ο Υπουργό μου απευθύνε δύο επιστολέ, τι οποίε έχω διανύμει και στα μέλη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, στι οποίε μα έδωσε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τι παράνομε διελεύσει, ε, του χώρου υποδοχή, ε, τι διαδικασίε παροχή ασύλου, τη ένταξη των ε, μεταναστών και έτσι έχει διατηρηθεί μεταξύ μας επικοινωνία όπως και τον Ιούνιο. Ελπίζω σε μία ακόμη σήμερα ε, εντελεχή ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βίτσα σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες ε, και τα διδάγματα που μπορούμε να αντιλήσουμε από την ελληνική εμπειρία ε, και το θέμα της μεταναστευτικής ροής σήμερα, πώς εξελίσσεται η κατάσταση, καθώς επίσης και ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε και συζητήθηκε και στο Συμβούλιο Στερικών ε, Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα, το ζήτημα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και πώς εφαρμόζεται. Και στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε τη δική του δουλειά, έχει εγκρίνει την εντόλη για το Δουβλίνο. Είμαστε όμως σε αρκετά δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, διότι εμείς κάναμε τη δουλειά μας πάνω σε διάφορους φακέλους που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, όμως όπως είδατε και στο Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, ε, είμαστε σε πολύ ε, δυσχερή θέση καθότι ζητείτε το πακέτο αυτό, αυτή η δέσμη μέτρων να κατατμηθεί σε διαφορετικά ε, κομμάτια. Αυτό θα ακούσω και τη δική σας άποψη. Επίσης, ό,τι αφορά τα προσωρινά μέσα, στις τις προσωρινές ρυθμίσεις, ε, ποια είναι η δική σας άποψη, εν και μιας πιο ε, οριστικής διευθέτησης, ήθελα θα ακούσω τη δική σας προοπτική και την άποψη των συναδέλφων βέβαια. Έχουμε καλέσει μέλη και της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ως Επιτροπή. Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι κατάφεραν να είναι εδώ γιατί ζητήσαμε να είναι ανοιχτή και προς αυτούς η σημερινή μας συνεδρία γιατί τους ενδιαφέρουν ε, το, το τι γίνεται και με τους καταβλισμούς ε, προσφύγων κυρία Μακάβαν και εγώ προσωπικά επισκεφθήκαμε και τα νησιά με τη συνεργασία της κυβέρνησης στην οποία είμαστε ευγνώμονες. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό, αφού τον ευχαριστήσω εκ νέου για την παρουσία του εδώ και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ε, good morning to everyone. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε και κύριοι. Θα συνεχίσω στα ελληνικά, όμως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορώ για δεύτερη φορά να είμαι εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και να σας ενημερώσω και να συζητήσω μαζί σας για την κατάσταση και τις προσπάθειες που καταβάλουμε εν ώψη και των δυσκολιών για τη διαχείριση λοιπόν το δυσκολίων στο προσφυγικό μεταναστευτικό και για την ευρωπαϊκή διαχείριση του θέματος και το νέο κανονισμό για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το αποκαλούμε. Και τώρα περνώ στα ελληνικά. Επειδή και στα ελληνικά είναι η ομιλία μου, οπότε θα δυσκολευτώ να τον μεταφράζω. 2018 βρίσκονταν στην Ελλάδα πάνω από 70.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Κατά το 2018 εισήλθαν στην επικράτεια της χώρας 47.929 άτομα, από τα οποία 32.115 στα νησιά και 15.814 στα χερσαία σύνορα μέσω του ποταμού Εύρου. Ε, το 2017 είχαν εισέλθει στη χώρα και από τα, στα νησιά και στα ε, χερσαία σύνορα 34.707. Η αύξηση των εισρωών ε, το 2018 στραμμένη μεν νησιά ήταν της τάξης του 10% και σημειώθηκε κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο, ενώ στα χερσαία σύνορα ήταν 284%, δηλαδή το 2017 είχαμε 5.500 αφήξεις, το 2018 15.814 αφήξεις. Στο τέλος του 2018 βρίσκονταν στα νησιά 14.615 άτομα, εκ των οποίων 11.683 στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και τα υπόλοιπα φιλοξενούνται είτε σε διαμερίσματα, περίπου 1.400 άτομα, είτε ε, και αυτό γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία, που διαχειρίζεται η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες ε, με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε στη δομή φιλοξενίας Καρατεπέ, ένα κέντρο φιλοξενίας στη Λέσβο, το οποίο έχει περίπου 1.000 άτομα, 1.150 άτομα. Η πρώτη και κύρια έγνοια μας το 2018 ήταν η όσο το δυνατόν άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρθηκαν από τα νησιά σε εποπτευόμενες από το κράτος δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα 29.090 άτομα, στα οποία είτε έχει χορηγηθεί καθεστώς προστασίας ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με βάση το πρωτόκολλο ευαλωτότητας. Πιο συγκεκριμένα, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν 14.887, από τη Σάμο 5.611, από τη Χίο 5.031, από την Κο 1.724, από τη Λέρο 1.330 και από τα άλλα τα νησιά 507 άτομα. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η παρουσία μας στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγαίου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι συνεχής σε επιχειρήσεις διάσωσης ε, τόσο από το λιμενικό όσο και από το πολεμικό ναυτικό με αποτέλεσμα να έχουν σωθεί χιλιάδες άνθρωποι από βέβαιο πνιγμό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι θάνατοι που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας κατά κύριο λόγο, δηλαδή το 90% προέρχονται από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Οι δε θάνατοι είναι περίπου 38, εκ των οποίων οι 20 είναι στην Εθνική Οδό της Εγνατίας. Ε, πνιγμούς είχαμε τέσσερις, τέσσερις σε ένα ατύχημα ε, στη Σάμο και σε ένα ατύχημα στον Εύρο. Ως πρώτην ενδοχό, βεβαίως όταν ε, ε, οι αριθμοί είναι αριθμοί. Ε, γιατί μια ζωή όταν χάνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και δεν είναι μόνο να συζητάμε σαν τους, αρι, ε, αριθμούς ότι εμείς έχουμε λίγους, κάποιοι άλλοι έχουν πολλούς. Κάθε άνθρωπος που χάνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ως προς την ενδοχώρα, στο τέλος του 2018, σε εποπτευόμενες από το κράτος δομές, διέμβαιναν με βάση το πρόγραμμα εστία σε διαμερίσματα 22.686 άτομα και στα 26 κέντρα φιλοξενίας που έχουμε στην ενδοχώρα 18.369 άτομα. Από τον Νοέμβριο δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε ξενοδοχεία και άλλα καταλήμματα όπου διαμένουν 6.793 άτομα. Ε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2018 έφυγαν από την Ελλάδα 6.782 άτομα. 322 στο πλαίσιο της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, 1.004 με βάση τις οικειοθελείς αποχωρήσεις στο πρόγραμμα που υποστηρίζει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και 5.456 άτομα μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των οικογενειακών επανενώσεων του υφιστάμενου καμονονισμού Δουβλίνου. Ως προς το άσυλο, το 2018 καταγράφηκαν 66.970 αιτήσεις ασύλου, ενώ το 2017 είχαν καταγραφεί 58.642. Είχαμε δηλαδή μια αύξηση περίπου 14% και έτσι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των, κρατών μελών στις αιτήσει ασύλου κατά κεφαλή, αμέσως μετά την Κύπρο, η οποία έχει ένα μικρό αριθμό αλλά μεγάλο σε σχέση με τον πληθυσμό της και τρίτη σε απόλυτους αριθμούς μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ως προς τις υπηκότητες των ετούντων άσυλων, ε, σημειώθηκε μείωση στις αιτήσει Σύριων, δηλαδή από 16.398 το 17 σε 13.390 αιτήσει το 18 και αύξηση στις αιτήσει των Αφγανών ε, από 7.566 το 17 σε 11.926 ε, το 18 και των Ιρακινών από 7.920 αιτήσει σε 9.731 αιτήσει. Ε, δηλαδή στην παρούσα φάση δεν έχουμε βασικά ροές καταγωμένων από τη Συρία, αλλά ροές καταγωμένων από το Αφγανιστάν, είτε αυτοί διαμένουν στο Αφγανιστάν ή διέμεναν στο Αφγανιστάν, είτε είναι Αφγανοί ε, οι οποίοι διέμεναν στο Ιράν. Συγχρόνως συνεχίστηκε η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για το άσυλο που υιοθετήσαμε το Μάιο του 2018 με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου. Αυξήσαμε κατά 25% τις αποφάσεις στη διαδικασία συνόρων στα νησιά και 50% στις επιδόσεις αποφάσεων στον πρώτο βαθμό. Επίσης, δημιουργήσαμε 8 επιπλέον επιτροπές προσφυγών με επιχειρησιακή έμφαση στα νησιά του Αιγαίου, άρα αυτή τη στιγμή έχουμε 20 επιτροπές προσφυγών και μειώθηκε ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων προσφυγών στα νησιά από την κατάθεση της προσφυγής από τις 124 μέρες στις 68 μέρες. Στις προσπάθειές μας για τη βελτίωση των υποδομών υποδοχής εντάσσεται και η μετεγκατάσταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΣΑΜΟ σε νέο σημείο του νησιού, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρατηρούνται στο υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το οποίο είναι το χειρότερο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και στην Ελλάδα, ε, δηλαδή είναι ε, ένα overcrowded ε, κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και είναι πρώτη μας προτεραιότητα να μειώσουμε τον ε, αριθμό. Ξέρουμε που είναι οι αιτίε, ε, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα ε, μόνο από τις τρεις τελευταίες μέρες. Πριν δύο μέρες έφυγαν από τη, από τη Σάμο για την ενδοχώρα 96 άτομα ε, οι οποίοι ήταν ευάλωτοι ή πήραν άσυλο. Εχθές το πρωί έφτασαν στην ε, Σάμο 103 ε, άτομα μετά από 4-5 μέρες που κανένας δεν έφευγε, κανένας δεν ερχόταν. Στη Σάμο θα δημιουργήσουμε ένα νέο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης 6 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα του νησιού, δυναμικότητας 1.200 ατόμων, ενώ το υπάρχον κέντρο θα κλείσει. Αυτό σημαίνει πως ο πληθυσμός στο κέντρο υποδοχής της ΆΜΟ θα πρέπει να μειωθεί κατά 2.500 ε, πολίτες τρίτων χωρών που είναι σήμερα, συν τον αριθμό των νέων αφήξεων. Το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή όλοι έχουν τον αριθμό ε, με το οποίο μπορούν να πηγαίνουν στα ιατρικά κέντρα και στα νοσοκομεία. Όλοι οι ανήλικοι έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα και είναι χαρακτηριστικό και πολύ καλό το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κανένα κρούσμα γρήπης μεταξύ του προσφυγικού μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Επίσης, τον Φεβρουάριο ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 300 γιατρών, ε, οι οποίοι θα διατεθούν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα κέντρα φιλοξενίας. Άρα ελπίζουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που μας τυραννάει πάρα πολύ καιρό, ιδιαίτερα στις διαδικασία ευαλωτότητας. Ω προ την εκπαίδευση των ανηλίκων, για τη σχολική χρονιά 2018-2019, 12.500 παιδιά παρακολουθούν μαθήματα στα δημόσια σχολεία ή σε δομές ε, υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων. Συγχρόνως, σε κάθε κέντρο φιλοξενίας, αλλά και στα κέντρα υποδοχής με τελευταίο της άμμου, προσπαθούμε να λειτουργούν νηπιαγωγεία και τα έχουμε καταφέρει. Ως προς την ένταξη, εντείνουμε τις προσπάθειες για την εφαρμογή της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ενσωμάτωση που βασίζεται στην προσέγγιση ότι η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων είναι αποτελεσματικότερη στο τοπικό επίπεδο. ω εκ τούτου, προβλέπει η Εθνική Στρατηγική τη συνεργασία και την εμπλοκή όλων των επιπέδων της διακυβέρνησης, κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και την εμπλοκή άλλων δρόντων όπως οι διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και του ιδιωτικού τομέα των τοπικών κοινωνιών στην εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης ολοκληρωμένης ένταξης, το οποίο το ονομάσαμε «Ήλιος», σε συνεργασία με το ΙΝΙΠΑΤΗ Αρμοστία και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στους Δήμους Στίβα και Λιβαδιάς, από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, ε, είχε εξαιρετική επιτυχία και τώρα προχωράμε αυτό το πρόγραμμα να το επεκτείνουμε σε δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, στοχεύοντας σε διάρκεια 12 μηνών να έχει ε, συμπεριλάβει 10.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στέγαση σε 5.000 άτομα για μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ένταξης. Ε, οι κύριοι πυλώνες του προγράμματος είναι μαθήματα ένταξης που θα περιλαμβάνουν εκμάθηση γλωσσών, ελληνική και αγγλική κατά κύριο λόγο, πολιτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό, δεξιότητες ζωής, αυτό είναι το πρώτο, δεύτερο καταγραφή των δεξιοτήτων και τρίτο στέγαση και χρηματική βοήθεια. Γενικά, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δικαιούχων ώστε να τους επιτρέψει να επανεισαχθούν σταδιακά στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ομαλή και μετάξυ ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον έχουν σχεδιαστεί σε κεντρικό επίπεδο προγράμματα για την ενσωμάτωση, η εφαρμογή των οποίων θα επικεντρωθεί και ήδη επικεντρώνεται σε μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για τους ετούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μετανάστες, το πρόγραμμα αυτά θα ωφελήσει 15.000 άτομα σε διάρκεια τριών ετών ε, που έχει μέσα και κατάρτιση και εξέβρεση εργασίες στον αγροτικό τομέα για 2.000 δικαιούχους και κατάρτιση και εξέβρεση εργασίας στον τουριστικό τομέα μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για 3.000 δικαιούχους διεθνούς προστασίας και βέβαια την καταγραφή δεξιοτήτων των ετούντων άσυλων. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι φανερό ότι δεν τα έχουμε λύσει όλα και ότι έχουμε πολλά προβλήματα γιατί είναι ένα, το μεταναστευτικό είναι ένα τελείως, μια τελείως δυναμική κατάσταση και εξαρτάται πάρα πολλές φορές και από τις ροές που έχουμε αλλά και με, από το τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την, το αίσθημα αλληλεγγύης και ανάληψης της συνευθύνης. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη βάση των κοινών μας αξιών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών. Είναι σαφές για μας ότι απέχουμε πολύ από αυτό το στόχο, καθώς δεν αντιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ευρώπης και όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Κάθε άλλο θα έλεγα. Ποιος είναι αυτός ο στόχος. Τίποτα λιγότερο από μια θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Δυστυχώς και παρά τις επίμονες συζητήσεις, το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει σε κοινή θέση ως προς την αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ειδικότερα του κανονισμού του Δουβλίνου. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταθέσει την πρότασή του για ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου ανθεκτικό στις μέλουσες προκλήσεις. Και είναι γνωστό ότι η ελληνική θέση συμφωνεί με, το, με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η Ελλάδα συγχρόνως με αυτό έχει επιδείξει επικοδομητικό πνεύμα στις διαπραγματεύσεις και έχει αποδεχθεί το κείμενο που διαμορφώθηκε επί Βουλγαρικής Προεδρίας σαν μια βάση για την έναρξη των τριλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να το πω ξανά, εμείς ε, ταυτιζόμαστε σχεδόν με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά συμβιβαζόστηκαμε στην πρόταση της Βουλγαρικής Προεδρίας για να αρχίσουν οι τρίλογοι. Αυτό βέβαια δεν το αποδέχονται μια σειρά χώρες και αυτό μας δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Παρά την αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης στην Ανατολική και Δυτική Οδό της Μεσογείου, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ επιμερισμού ευθυνών και αλληλεγγύης που θα ελαφρύνει τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής που βρίσκονται σε συνεχή πίεση. Όμως, δεν πρέπει να παραμείνουμε ως Ευρώπη, ως κράτη-μέλη, όμοιροι των εσωτερικών πολιτικών επιδιώξεων ορισμένων κρατών μελών ούτε να ανεχθούμε και να ανεχόμαστε ξενοφοβικές και ρατσιστικές προσεγγίσεις και πολιτικές. Είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα πριν τις ευρωεκλογές του Μαΐου προς τις κοινωνίες και την κοινή γνώμη των κρατών μελών πρώτης υποδοχής, ότι δηλαδή η Ευρώπη δεν μας έχει αφήσει μόνους να διαχειριστούμε τη μεταναστευτική πρόκληση. Η μη πρόοδος στην των διαπραγματεύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και ιδιαίτερα του κανονισμού του Βλήνου διευκολύνει κατά τη γνώμη μας τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης που τελικά αυτά αποφασίζουν ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει στην Ευρώπη. Οι επτά νομοθετικές προτάσεις της δέσμης ασύλου είναι αλληλένδετες και ως εκ τούτου πρέπει να υιοθετηθούν ως πακέτο ανεξαρτήτως στο σταδίου διαπραγμάτευσης που βρίσκεται η κάθε μία. Έως ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του κανονισμού του Βλήνου, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί με σαφές χρονοδιάγραμμα έως το Μάιο του 19 ένας μεταβατικός μηχανισμός αλληλεγγύης ή ειδικό ή ειδικά προγράμματα για κάθε χώρα πρώτης υποδοχής σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε χώρας που θα έχει έως αναπόσπαστο μέρος του την υποχρεωτική ανακατανομή ή μετεγκατάσταση. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί από τα κράτη-μέλη που είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν και με τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την Ελλάδα. Ο μεταβατικός αυτός μηχανισμός θα πρέπει να έχει τα εξής 7 βασικά σημεία. Πρώτο, ότι ο μεταβατικός μηχανισμός είναι καθαρό ότι αφορά στην εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Η έννοια της αλληλεγγύης είναι θεμελιώδης αρχή της Ένωσης και νομική υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που βρίσκονται σε πίεση. Και μου, μου θυμίζει αυτό το γεγονός ότι κάποια στιγμή μια χώρα, δεν θα πω το όνομά της, εκδηλώνοντας την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα το 2015 Έστειλε κασόνια, έστειλε κυβότια, γεμάτα ε, μαχαίρια και πυρούνια. Ε, έχουμε στην Ελλάδα μαχαίρια και πυρούνια, άλλα πράγματα ε, χρειαζόμαστε. Δεν ήταν το κύριο δηλαδή αυτό. Άρα όταν κάνεις αλληλεγγύη, την κάνεις στη βάση των αναγκών που έχει αυτός που θέλει την αλληλεγγύη. Και την αλληλεγγύη τη θέλουν δύο. Πρώτο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και δεύτερο το χρειάζονται, τη, χρειάζονται ε, οι χώρες πρώτης υποδοχής. Ως προς την εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης, δηλαδή το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι ανταλλάξιμη με τις κοινέ υποχρεώσεις φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα μέτρα στήριξης τρίτων χωρών. Το δεύτερο από τα 7. Αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού θα πρέπει να είναι ο επιμερισμός της ευθύνης δηλαδή ο υποχρεωτικός επιμερισμός των ετούντων άσυλο στις χώρες οι οποίες θα μπουν σε αυτό το ε, σύστημα. Το τρίτο, ο μηχανισμός θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλες ανεξαιρέτως τι μεταναστευτικές οδούς, δηλαδή και στην Ανατολική και στην Κεντρική και στη Δυτική Μεσόγειο. Γιατί ένας μεταβατικός μηχανισμός που έχει αυτή τη στιγμή ε, προταθεί από τη Γερμανία και τη Γαλλία αφορά κατά κύριο λόγο την Κεντρική Μεσόγειο, ε, δηλαδή περισσότερο τις περιπτώσεις που αφορούν την Ιταλία και την Ισπανία. Τέταρτο, τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν θα συμμετέχουν εθελοντικά στο μηχανισμό. Αλλά από τη στιγμή που θα συμμετέχουν εθελοντικά, οι δεσμεύσεις του μηχανισμού θα είναι υποχρεωτικές. Το πέμπτο, το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος, δηλαδή το μέγιστο των δυνατοτήτων κάθε κράτους μέλους, θα πρέπει να οριστεί αντικειμενικά σύμφωνα με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό που έχει το κράτος μέλος. Το έκτο, με τον τρόπο αυτό όλα τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν στο μηχανισμό, που θα συμμετέχουν στο μηχανισμό, θα συμμετέχουν εξίσου στον επιμερισμό των ευθυνών ως προς την υποδοχή, την εξέταση ετοιμάτων ασύλου, την ενσωμάτωση των δικαιούχων, την προστασία και την επιστροφή των μη δικαιούχων. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια επαρκή στήριξη από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και απαραίτητη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με μία έννοια επιμένουμε ότι όσα κράτη-μέλη θέλουν να συμμετάσχουν ε, στο μηχανισμό θα πρέπει να βοηθηθούν και μέσα από μια σειρά διαδικασίες τα κράτη-μέλη που δεν θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν κάποιες ποινές. Επιτρέψτε μου μια σημείωση, επειδή αρκετοί έχουν θέσει το θέμα του διαχωρισμού, το screening δηλαδή, μεταξύ προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο του μεταβατικού μηχανισμού. Δεν υπάρχει ορισμός screening σε επίπεδο Ένωση και ω εκ τούτου θα πρέπει να οριστεί ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσει και πολλαπλές ερμηνείε. Η Ελλάδα θεωρεί ότι η εξέταση μια αίτησης επί του παραδεκτού ή επί της ουσίας δεν αποτελεί screening, αλλά πλήρη εξέταση της αίτηση. Περαιτέρω, θα πρέπει να διασφαλιστεί αν αυτό περάσει η αντικειμενικότητα της διαδικασίας και ποιος θα φέρνει την ευθύνη του διαχωρισμού. Δηλαδή θα, τον φέρει, θα τη φέρνει το κράτος μέλος, θα, το φέρει, θα τη φέρνει η ύπατη αρμοστία, ποιος τέλος πάντων θα έχει αυτή την, ε, τη διαδικασία. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή αντίληψη μεταξύ των κρατών μελών για το ποιος δικαιούται διεθνούς προστασία με εναρμόδυνση του προσφυγικού προφίλ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χάνονται άνθρωποι στη Μεσόγειο και στις ερήμους της Βόρειας Αφρικής. Παρά τη συντριπτική μείωση των προσφυγικών ροών, υπάρχουν μεταναστευτικές ροές που επιμένουν γιατί επιμένει η εξαντλητική φτώχεια αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είμαι πεισμένος πως το αντίδοτο στην παράτυπη μετανάστευση και στη διακίνηση ανθρώπων είναι η βοήθεια στις χώρες καταγωγής αλλά και η νόμιμη μετανάστευση. Στο Μαρακές η ανθρωπότητα έκανε ένα πρώτο βήμα. Χρειάζεται να συνεχίσουμε. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτη και ανθρώπινη νομοθεσία για τη μετανάστευση και ασίγαστη καταδίωξη των εγκληματικών συμμοριών και οργανωμένων συμφερόντων διακίνησης ανθρώπων. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την παρέμβασή μου με κάποιες σκέψεις εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών. Δεν είναι η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή σα και να συζητήσουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στι μέρε μα και ιδιαίτερα στο με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και κάθε φορά, με κάθε ευκαιρία, θέλω να τονίσω την κεντρική σημασία που έχει η δημοκρατία, η λογοδοσία, η λαϊκή νομιμοποίηση όλου του θεσμικού συστήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρώπη πέρασε μια δεκαετία που έφερε στην επιφάνεια προβλήματα και ατέλειες στο οικοδόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε κρίση θεσμική, κρίση βαθιά πολιτική. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα κεντρικό ζήτημα που θα κυριαρχήσει στην προεκλογική περίοδο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις εκλογές, ευρωεκλογές τον Μάιο. Άρα θέλω να απευθύνω από αυτό το βήμα έκκληση μέσα από εσά τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν πρέπει να επιτρέψουν να επικρατήσουν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, οι δυνάμεις που προωθούν εθνικές επιδιώξεις αντί ευρωπαϊκών πολιτικών και προσεγγίσεων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη να υπερασπιζόμαστε τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες που αποτελούν τη βάση του κοινού μας οικοδομήματος. Από την πλευρά μου ευελπιστώ στη συνέχιση της καλής συνεργασίες μας με το Ευρωκοινοβούλιο, τη δημοκρατική δηλαδή φωνή των Ευρωπαίων πολιτών. Εσιοδοξώ ότι και μετά τις ευρωεκλογέ θα συνεχίσουμε την προσπάθεια στην εξέβρεση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων για τα κοινά μας προβλήματα στη βάση της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας. Σε μια κατεύθυνση που θα αξίζει πραγματικά να λέγεται ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βίτσα. Πολλά στοιχεία μας δώσατε σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και σχετικά με το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα ΣΥΛΟΥ και την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους Ευρωβουλευτές εάν έχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Σπινέλη, παρακαλώ. Thank σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τον Έλληνα Υπουργό ε, για την επίσκεψή του τούτη στην Επιτροπή μας, για την συνεχή παρουσία του στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να οργανώσουμε συναντήσεις και με άλλες χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να εξετάσουμε τις μεταναστευτικές πολιτικές. Σκέφτομαι ιδιαίτερα ε, τις χώρες με προβληματική πολιτική, όπως είναι η Ιταλία. Και χώρες με πολύ πιο προβληματικές πολιτικές από τη Ελλάς. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς τον Υπουργό όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου καθώς ε, και τις ε, προσωρινές ρυθμίσεις. Όσον αφορά λοιπόν τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις χώρες στην πρώτη γραμμή, ιδιαίτερα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Όσον αφορά τον προσωρινό μηχανισμό, την μεταβατική ρύθμιση, δεν είναι σαφές ότι θα αλλάξουν γνώμη όσοι είναι ε, κατά της μεταρρύθμισης του κανονισμού του Δουβλίνου. έχει προταθεί στο Συμβούλιο κατά τη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ακολουθεί την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό Δουβλίνο 3. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ, προτείνεται κάποιο είδους διευρυμένη συνεργασία. Αλλά αυτή η διευρυμένη συνεργασία ανάμεσα σε ποιους θα είναι και ποια θα είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του καθενός. Έχω επίσης μία ερώτηση σχετικά με τις όλο και περισσότερες άτυπες διμερείς ρυθμίσεις που βλέπουμε να εμφανίζονται ανάμεσα σε κράτη-μέλη σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Πολύ με ανησυχεί το θέμα αυτό. Μάλιστα έχουμε έκθεση έκρηση για ακριβώς αυτό το θέμα. Διότι η τάση είναι μάλλον απώλεια των εγγυήσεων που έχουμε στον ισχύοντα κανονισμό του Δουβλίνου. Φαίνεται να έχουμε οπισθοχώρηση και σε σχέση με τον κανονισμό Δουβλίνο 3. Επίσης έχει υποβληθεί μια ενοποιημένη έκθεση τον περασμένο Ιανουάριο που επισημαίνει την έλλειψη καταλημάτων. Επισημαίνεται επίσης ότι το σύστημα δεν λειτουργεί καλά για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα ήθελα λοιπόν ε, τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τη διαδικασία αυτή που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή σχετικά με το Δουβλίνο. Ναι, θα πρέπει να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι υπάρχει η συζήτηση για κατάργηση αυτής της δέσμης μέτρων. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τη δική σας άποψη, τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει. Θα ήταν ε, χρήσιμο. Η κυρία Βίξτρομ είναι η συγγήτρια για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Τη δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι είσαστε πολύ τολμηρός άνθρωπος. Τολμάτε ακόμα να μιλάτε για αλληλεγγύη, που δεν είναι η λέξη που συνήθως χρησιμοποιούμε εμείς που μιλάμε για τη μετανάστευση, διότι απλά συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σήμερα. Όχι στον τομέα της μετανάστευσης τουλάχιστον σε σχεδόν όλα τα άλλα θέματα, στην εσωτερική αγορά, την αλληλεία, τα χημικά, τα τρόφιμα, τα φάρμακα. Ε, κυριαρχεί η αλληλεγγύη. Στη μετανάστευση όμως δεν υπάρχει. Και έχουμε πολλές αποδείξεις γι' αυτό. Είσαστε λοιπόν πολύ θαραλέος άντρας που μιλάτε για αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη, μια πολύ όμορφη ελληνική λέξη. Θα ευχόμουν να ήταν δυνατό να μιλάμε για μετανάστευση στον τομέα, για ε, αλληλεγγύη, συγγνώμη, στον τομέα της μετανάστευσης. Και τα δύο τρίτα αυτού του κοινοβουλίου υπέγραψαν ε, ένα κείμενο που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για αλληλεγγύη στον τομέα της μετανάστευσης. Αλλά έχουν περάσει πολλοί μήνες και βρισκόμαστε σε κατάσταση πατ, διότι έχουμε πέντε ή έξι ε, χώρες που μπλοκάρουν την πρόοδο και ίσως όπως είπε η κυρία Σπινέλη και όπως αναφέρατε και εσείς αν και μάλλον δεν το είπατε πολύ ε, ξεκάθαρα μάλλον η διευρυμένη συνεργασία είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε και οι χώρες που δεν θα συμμετέχουν στις εργασίες αυτές, ε, αυτοί που δεν ε, συμμετέχουν ε, στις προσπάθειες υποδοχής, θα μπορούσαν ενδεχομένως να πληρώσουν για να απαλλαγούν. Θεωρείτε ότι αυτός είναι τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έτσι, θα μπορούσαμε ε, σήμερα που βλέπουμε πολύ μειωμένε εισρωές, ε, ήρθανε μόλις 95.000 ε, πέρσι, ενώ το 2015 ήρθαν 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να αναγκάσουμε τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς να μιλήσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο σύστημα. Παρότι βρισκόμαστε σε ιστορικά χαμηλό αυτή τη στιγμή, έξι άτομα πεθαίνουν καθημερινά στη Μεσόγειο. Κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κυριακή, Δευτέρα, κάθε μέρα, έξι εκατομμύρια άνθρωποι, έξι άτομα, χάνουν τη ζωή τους και έτσι χάνονται και οι ελπίδες για καλύτερο μέλλον στον μαζικό αυτόν τάφο στον οποίο έχει μετατραπεί η Μεσόγειος. Πιστεύετε λοιπόν ότι η διευρυμένη συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλη μέθοδο. Και δεύτερον, γνωρίζω ότι ακούγονται πολλά. Το Συμβούλιο δεν είναι και πολύ διαφανές, ε, γι' αυτό όλοι κάνουν υποθέσεις. Πολλοί υποθέτουν ότι η Ελλάς μπλοκάρει τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό το ότι μιλάτε και λέτε ότι η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης. Η Ελλάς συμβάλλει σε μια λύση, διότι αυτή είναι η Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι και στο Συμβούλιο να δείξετε ότι η Ελλάδα είναι συνεργάσιμος εταίρος και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τον Υπουργό να ε, υπερασπίζεται τον κανονισμό του Δουβλίνου την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριος Κύρκος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να υπενθυμίσω ότι ήταν πολύ σημαντικό η επίσκεψή σου και της κυρίας Μακάβαν στη Μόρια, ε, όχι μόνο γιατί είδατε από πρώτο χέρι τις συνθήκες που ζουν οι πρόσφυγές μας, αλλά γιατί δείξατε και στους ανθρώπους ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίπλα τους. Ε, κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Το ίδιο φιαλτικό μήνυμα βλέπουμε και σήμερα. Πρόσφυγε, οικονομικοί μετανάστες, άνθρωποι που ζητάνε άσυλο, περισσότεροι από αυτού που οι δομές φιλοξενίας και υποδοχή μπορούν να αντέξουν. Μια δήλωση με την Τουρκία που λειτουργεί στο Αιγαίο, αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε ότι η Τουρκία με τι τεράστιε πιέσει που δέχεται στι προσφυγικές τη ροέ και από την κοινωνική ένταση η οποία αυξάνει μεταξύ κατοίκων και μεταναστών θα συνεχίσει για πολύ καιρό να ε, κρατάει τα κλειδιά της, ε, του ευρωπαϊκού προβλήματος. Και η μετακίνηση από τα, από τα νησιά στην ενδοχώρα επιβαρύνονται και ολοκληρώνεται, καλύπτονται όλες οι δομές φιλοξενίας, τα προγράμματα ένταξης γονατίζουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για μια χώρα που βρίσκεται ακόμα, έστω και σε λιγότερο βαθμό, σε μια οικονομική κρίση. Και βλέπουμε πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές, που όπως σωστά είπε η κυρία Βίξτρομ δείχνουν δείγματα αλληλεγγύης, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες πολιτικές, είτε η ψηφιακή αγορά, είτε η κοινή εξωτερική πολιτική, είτε η οικονομική ολοκλήρωση, στο θέμα του προσφυγικού, όταν το ζήτημα σκάσει, θα είναι πάρα πολύ φανερό. Μπορούμε να μεταθέτουμε την, την οικονομική ολοκλήρωση για ένα, δύο, τρία χρόνια. Δεν θα βγουν οι άνθρωποι στον δρόμο από τράπεζε που κλείσαν. Αν η Ελλάδα σκάσει όμω, τα προβλήματα θα είναι, θα είναι μπροστά στα μάτια μα. Και σας ρωτάω, η ερώτησή μου σε εσά είναι, αν δεν ε, μπορέσουμε να περάσει η πρόταση του Κοινοβουλίου που είναι για την αναθεώρηση του Δουβλίνου, αν δεν προχωρήσει παρά τις συζητήσεις που γίνονται πολύ καιρό τώρα για αυτή την αυξημένη συνεργασία, αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως είναι, κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες. Πόσο καιρό θα κάνει η Ελλάδα, πόσο καιρό θα μπορέσει η Ελλάδα ακόμα να αντέξει και τι θα σημαίνει μια χώρα που δεν αντέχει να υποδέχεται άλλους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά εσείς που χειριζόσαστε αυτό το ζήτημα και τι σημαίνει και για την Ευρώπη αυτό. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Kirkos. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Κύρκο, η κυρία Στίβενς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τις απόψεις σας και τις εμπειρίες σας σχετικά με τον αντίκτυπο της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς έχει επηρεάσει την πρώτη γραμμή κρατών μελών η μεταρρύθμιση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. Πώς έχει επηρεαστεί η χώρα σας δηλαδή ως κύριος προορισμός πολλών μεταναστών. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουμε την αρχή της ασφαλούς χώρας προέλευσης και της ασφαλούς χώρας διέλευσης. Οι κανόνες λοιπόν λένε ότι οι αιτήσει ε, μεταναστών από για παράδειγμα την Τουρκία μπορούν πολύ γρήγορα να διεκπεραιωθούν για να διευκολυνθεί η γρήγορη επιστροφή των ε, παράνομων μεταναστών. Έχουμε δηλαδή μια διαδικασία fast track. Οι αρχές αυτές ενσωματώθηκαν ε, στην ελληνική νομοθεσία, ε, εφαρμόζοντας έτσι τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και αυτή η διαδικασία fast track έχει επηρεάσει τις αφήξεις και προτείνεται και σε άλλα κυρίαρχα κράτη να ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση, δηλαδή να συνάψουν συμφωνία σε επανεισδοχή με άλλες χώρες της Μεσογείου, ώστε να διευκολυνθεί η γρήγορη επιστροφή τους μετά από ε, γρήγορη εξέταση των αιτήσεών τους. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι πιο σύντομη. Πόσοι μετανάστες επεστράφησαν στην Τουρκία σύμφωνα με τη συμφωνία από την Ελλάδα και γιατί είναι τόσο χαμηλό ο αριθμός αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την απάντησή σα. Η κυρία Κουτσίσκα, παρακαλώ. E, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας συγχαρώ, διότι βλέπω ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει όλο και καλύτερα με τις ε, μεταναστευτικές ροές, που βέβαια μειώνονται κιόλας, ε, οπότε αυτό απλοποιεί κάπως ε, την κατάσταση. Και εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η κατάσταση στο Συμβούλιο η ιδέα δηλαδή διάσπασης της δέσμης μέτρων του Δουβλίνου, η διάσπαση της, του πακέτου αυτού, το ερώτημά μου προς εσάς κύριε Υπουργέ είναι ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν και τι δυνατότητες ή πιθανότητες υπάρχουν να παραμείνει το πακέτο ως έχει. Υπάρχουν πιθανότητες και πόσες είναι αυτές. Δεύτερο ερώτημα. Είπατε κύριε Υπουργέ ότι θα πρέπει να αναλάβει δράση η Frontex και αν σας κατάλαβα καλά πρέπει να εννοείται να δράσει καλύτερα η Frontex. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η δράση της Frontex. Θα ήθελα να τις μοιραστείτε μαζί μας, αν έχετε κάποιες προτάσεις. Και τελευταίο ερώτημα. Γνωρίζουμε πως η μεταναστευτική πίεση υποχωρεί, μειώνεται και για την Ελλάδα. Όμως, στη Μεθόριο, στον Εύρο, βλέπουμε να αυξάνεται η κίνηση. Γιατί, γιατί υπάρχουν περισσότερα άτομα τα οποία συγκεντρώνονται εκεί. Ευχαριστώ. Η καλύτερη ερώτηση ήταν αυτή. ποια κράτη ε, μέλη φταίνε, αλλά κάπως υποπτεύομαι ότι δεν θα πάρουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Τζούντιτ Σαρτζεντίνη τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Επιτροπή κατά των βασανιστήριων ε, δημοσιοποίησε μια έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και τους ετούντες άσυλο. και μιλάει για τα αστυνομικά τμήματα στα οποία κρατούνται για εβδομάδες ή και μήνες ε, οι μετανάστες. Ε, ένα τετραγωνικό μέτρο μπορεί να κινηθούν ε, και υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα. Δεν άκουσα όμως κάτι από εσάς κύριε Υπουργέ. Νομίζω όμως θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να μας αναφέρετε κάτι πάνω σε αυτή την έκθεση της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, Τζούντιτ. Κυρία Σίντο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω. Λέγομαι Μιχαήλα Σόιντροβα. Πριν 14 ημέρες ε, ξαναειδωθήκαμε και πραγματικά σας είμαι ευγνώμων γιατί φερώσατε χρόνο ε, και με συναντήσατε. Γνωρίζετε την πρωτοβουλία ε, της οποίας είχουμε εκ μέρους της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το αφήνω όμως κατά μέρος αυτό και θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα από τα δικά σας ε, ε, μηνύματα, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες αυτών οι οποίοι εργάζονται επί τόπου. Αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή που εργάζονται με τα παιδιά, με τις οικογένειες ε, που με μεγάλο επαγγελματισμό φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται για εθελοντές ε, οι οποίοι καλωσορίζουν τους μετανάστες αυτέ αυτούς. Ξέρω ότι υπάρχει μια μακρά διαδικασία από την άφηξη των μεταναστών μέχρι τη δεκπεραίωση των αιτήσεών τους και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν λόγοι για αυτή την καθυστέρηση. Όμως ε, οι άνθρωποι αυτοί ε, μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Βρίσκονται σε μια μετέωρη κατάσταση και πολλοί ε, τελικά αποφασίζουν χωρίς να περιμένουν την έκβαση της αίτηση να φύγουν και να προχωρήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα και πράγματι ε, στον Εύρο αυξάνονται οι αριθμοί. Το έχω ακούσει και εγώ. Δύο με πέντε χιλιάδες άκουσα. Άνθρωποι διέρχονται του συνόρου αυτού κάθε εβδομάδα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ψηλός αυτός ο αριθμός. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας ε, εκτιμήσεις. Αν έχουμε 2.000 μάλλον 200-500 ε, το μήνα, φτάνουμε στους 2.000 τη βδομάδα, φτάνουμε στους 2.000 το μήνα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται και με την ε, διεθνή προστασία. Δεν νομίζω ότι έρχονται από την Ερυθρότητα, από τη Συρία ε, οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πώς επαναπατρίζουμε αυτά τα άτομα, αυτούς τους ανθρώπους. Και σε ό,τι αφορά κάποια σχόλια των προλαϊσάντων συναδέλφων γνωρίζουμε ότι στα κράτη-μέλη αυξάνονται οι φωνές που λένε να βοηθήσουμε εκεί που οξύνονται τα προβλήματα, φτώχεια, βία, εκεί να βοηθήσουμε, σε αυτές τις περιφέρειες. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου, καλώντας, εποδεχόμενοι όλους ε, ε τους ε, ανθρώπους που φεύγουν από αυτές τις περιοχές του κόσμου. Πρέπει να βοηθήσουμε πιο με προτεραιότητα αυτούς που γνήσια χρειάζονται βοήθεια και αυτό δυσχεραίνεται. Υπάρχουν πολλοί οποίοι φεύγουν λόγω πολέμου, λόγω θρησκευτικής δίωξης και θέλουμε να έχουμε τις δυνατότητες να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς ακριβώς τους μετανάστες κατά προτεραιότητα. Αν βλέπουμε όμως μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας αυτόματα, ε, δυνάμει της Γενέβης, όταν αυτοί οι άνθρωποι ε, πολλαπλασιάζονται, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα που άμεσα χρήζουν ε, προστασίας και βοήθειας. Και έρχομαι στο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών των ασυνόδευτων ανηλίκων. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ελλάδα να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία που ήδη υπάρχει και όσοι ενδιαφέρονται είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν στην Τσεχική Δημοκρατία για παράδειγμα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα. Σας ευχαριστώ πάντως γιατί ξέρω ότι κάνετε το μέχρι το δυνατός λαός. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος άλλος, ε, ξέχασα κανέναν μήπως. Κύριε Υπουργέ, ήρθατε σε πολύ καλή χρονική στιγμή. Οι βουλευτές ενδιαφέρονται, όπως καταλαβαίνετε, για την κατάσταση. Πάντοτε θα μας ενδιαφέρει η κατάσταση ε, που ε, είναι γεμάτη προκλήσεις, γι' αυτό και θέλουμε να έχουμε ένα τακτικό ρυθμό ενημέρωσης πληροφόρησης, εξού και σας ε, προσκάλεσαμε για δεύτερη φορά, αλλά και από πολιτικές πλευράς αυτή η χρονική στιγμή είναι ενδιαφέρουσα λόγω του Δουβλίνου, λόγω της τάσης του Συμβουλίου. Παρακαλώ λοιπόν να σας δίνω ξανά το λόγο για να απαντήσετε στα ερώτημα των συναδέλφων. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις θα έλεγα ότι θα τις χωρίσω, τις, τις απαντήσεις μου να τις χωρίσω σε δύο μεγάλα κομμάτια. Το ένα κομμάτι αφορά το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και σε επίπεδο Συμβουλίου και το άλλο ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό προσφυγικό που έχουν όμως και ένα πιο πρακτικό ή νομικό ε, χαρακτήρα. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Συζητάμε για την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο περίπου δύο χρόνια. Περίπου δύο χρόνια, ίσως και παραπάνω. Γιατί το Δουβλίνο 3 κατέρευσε το 2015. Κατέρευσε, δηλαδή δεν εφαρμόστηκε καν. Ε, δύο χρόνια τώρα που συζητάμε, ε, κάθε φορά κάποια χώρα βρίσκεται ε, και ή κάποια ομάδα χωρών, κατά κύριο λόγο οι χώρες του Βίζαγκραντ, δεν φοβάμαι να τα πω γιατί τα λέω και με τους ε, συναδέλφους μας, οι οποίες μπλοκάρουν ακόμα και προτάσεις που, θα το πω όπως το λέμε στην Ελλάδα, βρε αδελφέ, δεν είναι για καμιά φοβερή τομή. Δηλαδή, η πρόταση της Βουλγαρίας, τι λέει, ότι όταν μια χώρα ξεπεράσει το capacity που έχει στην εξέταση ασύλου, δηλαδή 140, και ξεπεράσει το 140% τότε γίνονται δύο ψηφοφορίες ώστε να υπάρξουν περιπτώσεις που θα μεταφερθεί το αίτημα του ασύλου σε άλλη χώρα. Και στη μία ε, είναι η ψηφοφορία θετική και μετά από 15 μέρες είναι με αρνητική ψήφο, ε, δηλαδή αν δεν συγκεντρώσει αρνητικές και προχωράει η πρόταση της Επιτροπής και δεν γίνεται δεκτό. Δεν γίνεται δεκτό. Αφού βάζει κιόλα η Βουλγαρία, η Βουλγαρική Προεδρία, ε, πολλά βολοντάρι, πολλά εθελοντικά μέσα. Γι' αυτό λέω ότι εμείς είμαστε ε, με την ε, πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάζει μια υποχρεωτικότητα στη συνευθύνη και στην αλληλεγγύη. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη αλληλεγγύη και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος η αλληλεγγύη θα κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όποιος νομίζει ότι με τα τουφέκια ή με τα όπλα μπορεί να διατηρήσει απ' έξω ε, από την ε, Ευρώπη ανθρώπους οι οποίοι θα πεθάνουν στη χώρα τους και έρχονται στην Ευρώπη, τότε να έρθει να πάω να του δείξω μερικά μέρη στο Νεύρο. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει και αυτή ένα τείχος. Έχει φτιαχτεί τα παλιότερα χρόνια 12,5 χιλιόμετρα στο Νεύρο. Αν πάτε εκεί, θα δείτε ότι υπάρχουν ε, τζάκετ, ότι υπάρχουν γάντια, ότι υπάρχουν ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από πάνω από το τείχος. Τα βλέπουμε όμως και στην Αμερική καθημερινά αυτά τα πράγματα στα ε, ε, σύνορα ανάμεσα στι ΗΠΑ Αμερικής και Μεξικό. Άρα εγώ είμαι πεισμένο, αρκεί να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Αρκεί να μην υιοθετούμε την ατζέντα των ρατσιστών και των ξενοφοβικών για να πάρουμε περισσότερους ψήφους. Με αυτόν τον τρόπο δυναμώνουμε αυτές τις ομάδες. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου την, ε, γνώμη. Λέμε λοιπόν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια φοβερή στασιμότητα πάνω σε αυτό. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει στις τέσσερις από... τα τέσσερα από τα εφτά νομοθετήματα τα έχουμε συμφωνήσει. Πραγματικότητα είναι ότι τα έχουμε συμφωνήσει. Να προχωρήσουμε αυτά. Να κάνουμε split δηλαδή, να διαιρέσουμε και να, κάνουμε... να προχωρήσουμε αυτά. Ερχόμαστε εμείς σαν Ελλάδα και λέμε Μα συγχωρείτε, τα τέσσερα που έχουμε συμφωνήσει μέσα στο πακέτο είναι μόνο διασυνοριακές διαδικασίες. Border procedures. Δηλαδή, παίρνουμε τη μία διάσταση μόνο, μόνο τις διασυνοριακές διαδικασίες. Και στην ουσία, αν προχωρήσουμε τα τέσσερα, τότε η αναθεώρηση του μηχανισμού του όχι δεν πάει στις καλένδες, δεν θα γίνει ποτέ. Πολύ ωραία, νομίζω η κυρία Σπινέλη, δεν, θυμάμαι ποιος είπε, το, το εξή. Α, η, κυρία Βίξτρομ το είπε. Ε, ότι ε, ενώ σε όλα τα άλλα δείχνουμε ή σε πολλά από τα άλλα πιο σωστά, δείχνουμε αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεταναστευτικό καμία. Άρα στην ουσία με αυτόν τον τρόπο ευνοούνται οι χώρες που κρατάνε εθνική πολιτική. Μην με βάζετε τώρα να ονομάσω αυτές τις χώρες. Όμως κρατάνε εθνική πολιτική εις βάρος των χωρών της πρώτης υποδοχής. Μόνο αυτών. Όχι. Και εις βάρος των χωρών προορισμού. Δηλαδή ότι δεν παίρνει μία χώρα, το παίρνει τελικά και με διάφορους τρόπους, νόμιμους και παράτυπους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα καταμερισμού της ευθύνης και της αλληλεγγύης που θα διευκολύνει όλους. Αυτό είναι το, το βασικό. Γιατί μην μου πείτε ότι 100.000 άνθρωποι ή συνολικά 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από το 2015 δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στην Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τη στιγμή που η Ελλάδα των 10 ε, εκατομμυρίων φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 75.000 που έχουν έρθει από το 2015 και 550.000 που ζουν και έχουν ενσωματωθεί στην Ελλάδα από το, 1990 και μετά. Δηλαδή αυτή είναι η, η, η βασική μου σκέψη. Το ερώτημα όμως μπήκε ακόμα πιο έξυπνα. Ωραία και τι θα γίνει. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, δεν το έχω πει πουθενά, δεν το έχω πει ούτε στον Πρωθυπουργό της χώρας. Εγώ θα ψηφίσω θετικά ή θα ζητήσω η Ελλάδα να ψηφίσει θετικά σε οποιοδήποτε μηχανισμό θα μειώσει τους πνιγμούς στη Μεσόγειο. Δεν θα πάω να πω «Α, ξέρετε, εγώ χαλάω δικά μου λεφτά, της Ελλάδας δηλαδή τα λεφτά, στο λιμενικό, στο πολεμικό ναυτικό για να διασώζουμε ανθρώπους, ενώ οι άλλοι δεν χαλάνε και ότι πρέπει κάτι να πάρετε και από εμά. Θα το πω αυτό, αλλά δεν θα το δεν θα εκβιάσω με αυτό. Γιατί για μένα η ανθρώπινη ζωή, για μας η ανθρώπινη ζωή έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αλλά πρέπει να δούμε και κάποιε διαδικασίες δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα το αίσθημα τη και τη αλληλεγγύη και το δεύτερο το τιμωρητικό αίσθημα. Δηλαδή όταν θα πάμε να συζητήσουμε και θα το πω και σε εσά ανοιχτά. Το ε, επόμενο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για το 2021-2027, τότε εμείς θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις χώρες οι οποίες δεν συμβάλλουν στο μηχανισμό αλληλεγγύης, στο, πώς το λένε, στην, ε, στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό. Δεν θέλω να προχωρήσω ε, παρακάτω. Και εδώ δεν είναι ζήτημα χρημάτων. Δηλαδή έρχεται μια χώρα και λέει ε, «Α, εγώ θα δώσω λεφτά, αλλά δεν θα πάρω πρόσφυγες». Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι μοιραζόμαστε το βάρος. Η Ελλάδα κάνει πολύ περισσότερα και άλλες χώρες, δεν λέω, Δηλαδή, εμείς όλες τις προσωμιώσεις μπορούμε να εξετάζουμε 20 με 25 χιλιάδες αιτήσει ασύλου το χρόνο. Εξετάζουμε 66 χιλιάδες αυξήσεις το χρόνο. Εγώ σας το λέω και σας το προειδοποιώ. Βρισκόμαστε συνέχεια στο όριο ως υπηρεσίες ασύλου. Στο όριο. Και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους και τα λοιπά. Από αυτή την αδυναμία το να υπάρχει, όπως είπε η κυρία Σπινέλη, ε, ένα κοινό σύστημα ασύλου και ένα σύστημα συνευθύνης, αρχίζουν και βγαίνουν νέα φαινόμενα διαλυτικά κατά τη γνώμη μου για την Ευρώπη, δηλαδή να συνεχιστούν. Οι διμερείς συμφωνίες, για παράδειγμα. Οι εθνικές πολιτικές, για παράδειγμα. Για μας το βασικό και το κύριο είναι να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Επαναλαμβάνω, εμείς, σαν Ελλάδα, χωρίς να συμφωνούμε με την πρόταση της Βουλγαρικής Προεδρίας, την αποδεχτήκαμε σαν βάση για συζήτηση, ώστε να προχωρήσει ένα βήμα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το, το θα λέγαμε, ε, βασικό. Πολλοί λένε, λέει, ότι η Ελλάδα δεν αφήνει τις διαδικασίες να προχωρήσουν. Ποιες διαδικασίες δεν αφήνουμε να προχωρήσουν. Δεν αφήνουμε τις διαδικασίες οι οποίε επιτρέψτε μου να πω με το φίλο μου, το φίλο μου, πάντων με τον ε, συνάδελφό μου τον κύριο Κίρκλ, τσακωνόμασταν επί έξι μήνες ποιο είναι το κύριο. Αν το να, να πάμε στρατό στα σύνορα είναι το κύριο ή η συνθήκη της Γενέβης είναι το κύριο. Και λέμε τα, εύκολα αλλά τα μη παραδεκτά. Κάποιος που καταθέτει, κάποιος που καταθέτει αίτημα ασύλου έχει το δικαίωμα και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να του το αφαιρέσει να εξεταστεί αυτό το δικαίωμα, αυτό, αυτό το αίτημα. Δεν μπορεί κανείς να του το αφαιρέσει, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα. Το να βοηθήσουμε και να διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες από την Ευρώπη αυτό να γίνεται γρήγορα είναι ένα άλλο θέμα. Ή αν θέλετε είναι το βασικό θέμα. Είναι να δυναμώσουμε το ΕΑΖΟ, να έχουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου, να δυναμώσουμε τις υπηρεσίες μας. Σας είπα ότι στο δεύτερο επίπεδο στις προσφυγές εμείς καταφέραμε τις 124 μέρες να το πάμε στους 68. Έχει να κάνει βέβαια και με τις ροές, πόσες υποθέσεις έχεις, πώς μπορείς να... Άρα δεν είναι ότι δεν αφήνουμε τις διαδικασίες να προχωρήσουν. Δεν αφήνουμε μια πολιτική που επικεντρώνει μόνο στο στην ψευδεπίγραφη προστασία συνόρων και που θεωρεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εισβολής ε, όχι, δεν αφήνουμε να, να, προχωρήσει μια τέτοια λογική. Δεν αφήνουμε να προχωρήσει μια τέτοια λογική. Δεν είναι ούτε εισβολής, είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Επιστροφές. Το, από την Ελλάδα με βάση την κοινή δήλωση έγιναν 300 επιστροφές 310 ε, επιστροφές, το 2018 550 το 2017. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Με την έννοια ότι υπάρχει μια ολόκληρη νομική διαδικασία και βεβαίως υπάρχει και σωστά υπάρχει, η αρμοστία, διεθνής οργανισμός ε, μετανάστευσης, οι, συνήγοροι του πολίτη, οι ομπουσμαν δηλαδή, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, άνθρωποι ευαίσθητοι. Ε, ευαίσθητοι όχι με την έννοια της ευαισθησία που λέμε, αλλά ευαίσθητη σε επίπεδο των ε, ανθρώπινων ε, δικαιωμάτων, που εξαντλούμε την περίπτωση. Εξαντλούμε την περίπτωση πριν φτάσουμε σε αυτό. Εμείς στην Ελλάδα ακολουθούμε αυτή την πολιτική. Η πολιτική της έρευνας και διάσωσης και η, η πολιτική της φιλοξενίας με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και της εξάντλησης όλων των περιπτώσεων εξέτασης των ετοιμάτων ασύλου. Αυτό είναι το ε, βασικό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ε, ολοκληρώσω. Ε, με συγχωρείτε, αλλά μάλλον έγινε ένα λάθος. Εγώ δεν στην ομιλία μου, μάλλον το προηγούμενο κείμενο ήτανε, που το έκανα διορθώσεις, δεν μίλησα καθόλου για τη Frontex. Καθόλου για τη Frontex. Γιατί η υπόθεση της Frontex είναι μια υπόθεση που συζητιέται αυτή τη στιγμή και στη Σύνοδο των Υπουργών με πολλά νομικά ζητήματα, προβλήματα και με πολλά ζητήματα σε σχέση με το mandate της ε, Frontex. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω μόνο είναι ότι η Frontex θα πρέπει να ακολουθήσει την, ε, θα έλεγα, ε, εκείνο το κομμάτι του κανονισμού της που της λέει ότι πρέπει να ενεργοποιείται πάρα πολύ στο ζήτημα της έρευνας και διάσωσης στο σύντημα της έρευνας και διάσωσης. Εγώ, εγώ αυτό... Ε... Τώρα η τελευταία ερώτηση στην οποία θα απαντήσω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν ερωτήσεις... Α, σε σχέση με τα, τις κρατήσεις στα αστυνομικά τμήματα. Κοιτάξτε, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα κατά την περίοδο Απρίλιος, <clears throat> Αύγουστος, με τη μεγάλη αύξηση των ροών από τον Εύρο. Ε, αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι εχθές σε αστυνομικά τμήματα κρατούνταν στον Εύρο, κρατούνταν 90 άτομα σε όλα τα, ασφαλεια, τα αστυνομικά τμήματα ε, μαζί και πολύ γρήγορα προσπαθούμε να τους περνάμε. Αυτά τα 90 άτομα πριν τρεις μέρες δεν ήταν εκεί, ήταν κάποιοι άλλοι. Στο φυλάκιο όπου γίνεται η καταγραφή και μπορούν να φεύγουν. Νομίζω ότι η επικίνδυνη ερώτηση ήταν του Έλληνα Ευρωβουλευτή, του κ. Κύρκου. Ε, θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να φανταστώ ότι δεν θα βρεθεί καμία ευρωπαϊκή λύση. Ε, γιατί αν δεν βρεθεί καμία ευρωπαϊκή λύση, οι χώρες πρώτης υποδοχής και ιδιαίτερα η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ισπανία θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αυτό δεν θα το πληρώσουν μόνο αυτές οι χώρες, θα έλεγα θα το πληρώσει ολόκληρη η Ευρώπη. Ε, πώς θα γίνει αυτό, εγώ παλεύω να βρεθεί λύση. Δεν παλεύω να μην βρεθεί λύση. Αυτό είναι το ε, βασικό. Ε, και αυτό είναι το κεντρικό, αν θέλετε, πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι καθήκον μας είναι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση. Με βάση τις αρχές του διεθνού δικαίου, με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, με βάση τις πρώτες προσπάθειες στο Μαρακές, να βρούμε μια λύση. Ε, και από εκεί και πέρα καθήκον μας είναι να προσπαθούμε να βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις. Εμείς αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, να, να λύνουμε προβλήματα που υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την ε, διαμονή, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι τώρα είναι η Σάμος, πριν από πολύ καιρό, πριν από δύο χρόνια ήταν η Ιδωμένη, μετά ήταν ο Πειραιάς, μετά ήταν το Ελληνικό, το καλοκαίρι στις αρχές ήταν η Μόρια, τώρα δεν είναι η Μόρια. Ε, παλεύουμε για να τα λύσουμε. Τελείωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, uh, Minister. Κύριε Υπουργέ, ένα θερμό ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. και γνωρίζουμε όλοι ότι οι επαφές μας έχουν παραμείνει στενές ε, όλο αυτό το διάστημα που δοκιμάζεται η Ελλάδα, ιδίως στα νησιά της. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για την ενημέρωση και για το Δουβλίνο και για την πολιτική κατάσταση. Κύριε Σβίτσα, σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε μέλος της Επιτροπής σας, κάθε Ευρωβουλευτής ε, του Κοινοβουλίου είναι ευπρόσδεκτος να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά Παρακαλώ, μην έρθετε μόνο να επισκεφθείτε τη Μόρια, αλλά και τα άλλα κέντρα υποδοχής, τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και στην ενδοχώρα, αλλά και στα νησιά. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ ξανά, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Ετοιμάστε τις κάρτες ψηφοφορίας. 11 um, και 4 θα ψηφίσουμε. Um, Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι καθίστε για να ξεκινήσουν τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 11. 11 λέει ο πρόεδρος. 11 Πρόκειται για την ε, εκτελεστική απόφαση την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία, Μην ανησυχείτε. Αλλά καθίστε παρόλα αυτά. Έχουμε τον κανόνα 51 που ισχύει. Προτείνω να εγκριθεί έκθεση χωρίς τροπολογίες, εκτός εάν... Ευχαριστώ που κάνετε ησυχία, εκτός εάν φτάσουμε στον μέσο όρο 10% έξι βουλευτές δηλαδή να διαφωνήσουν. Υπάρχουν διαφωνίες, όχι. Επομένως η έκθεση εγκρίνεται. Εγκρίνεται και η έκθεση του κυρίου Σκρίπεκ. Συγχαρητήρια κύριε Σκρίπεκ, αν είστε εδώ. Περνάμε στο σημείο 12. Συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά έχω να διαβάσω εδώ διάφορα για το σημείο 12 που είναι η ρύθμιση με το βασίλειο της Νορβηγίας, τη δημοκρατία της Ισλανδίας. την Ελβετική Συνομοσπονδία και το πριγκιπάτο του Λίχτενστάιν όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ε, τεχνολογιών πληροφοριών μεγάλη κλίμακα στον χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Για μακρό. Όπω το σύστημα Ιουλή. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα έχουμε αυτό το νέο κανονισμό για το ίδιο Λίσα που προβλέπει την ολοκλήρωση των νέων διευθετήσεων, τις οποίες πρέπει να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν συμφωνήσει στις 27 Σεπτεμβρίου οι να ακολουθηθεί η απλουστευμένη διαδικασία το άρθρο 51. Κυρία Μακοβέη έχει αναλάβει το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Είναι εδώ κύριε Μακοβέη, δεν είναι. Ως πρόεδρος λοιπόν, να με το άρθρο 51 προτείνω να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες η έκθεση εκτός εάν φτάσουμε πάλι να έχουμε 10% 6 ε, μέλη δηλαδή που θα ενίστανται σε αυτή την πρόταση. Ε, υπάρχει κάποιος που ενίσταται? Όχι. Επομένως εγκρίνεται η έκθεση και συγχαίρω την κυρία Μακοβέη. Και τώρα Περνάμε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτο δικαίου και την καταπολέμηση τη διαφθοράς στην Ένωση, ιδίω Μάλτα και Σλοβακία. Η κυρία Ιντβελτ, η συγγήτρια. Θέλει το λόγο, μήπω σοφή πριν την ψηφοφορία. Όχι, άρα περνάμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία. And um, we go first of all to paragraph And the Παράγραφος 4. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. And that's also... Εγκρίνεται. Παράγραφος 21 με το συν Βουλγαρία. And Bulgaria. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 παράγραφος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τέλος, ονομαστική ψηφοφορία, η τελική, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται 40 ψήφοι πέρα, 7 κατά 6 αποχές, χαρητήρια στην εισηγήτρια. Προχωρούμε στην πρόταση απόφαση του Συμβουλίου, με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικού αγώνε και άλλε αθλητικέ διοργανώσει. Η Σιλβί Βον Κάφμαν, η συγγήτρια, θέλετε το λόγο. Α, δεν είναι καν εδώ, κυρία Κάφμαν. Δεν βλέπω, συγγνώμη, σήμερα δεν βλέπω. Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία που είναι μία και μόνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα άρχεται. Πέρας. Πέρας. Εγκρίθηκε 38 ψήφοι υπέρ ψήφι κατά μία αποχή. Συγχαρητήρι στη Σίλβια Ιβών. Και προχωρούμε στο σημείο 15 κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Έκθεση Μάμικινς. Ενοποιημένη πρόταση του αποτελέσματος των διοργανικών διαβουλεύσεων. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο ο εισηγητής. Ο Αντρέη όχι. Άρα περνάμε στην ενιαία αυτή στη μόνη ψηφοφορία άρχεται. Πέρας ψηφοφορία. Πάρα πολύ καλά. 52 ψήφοι, όλες υπέρ. Χαίρομαι που άξιζε τελικά όλος αυτός ο χρόνος ε, στη... στον τριμερή διάλογο. Εγώ δεν έχω πάντοτε την ίδια εμπειρία με τους τριμερείς διαλόγους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πού είναι, ποιο, ποιο είναι. Α, θέσπιση του Ταμείου Ιστορικής Ασφάλειας, η γήτρια η Μόνικα Χολμάιερ. Θέλει το λόγο η Μόνικα, όχι. Συμβιβαστική 16 που καλύπτει τις τροπολογίες 20 και 21 άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει είμαστε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 137 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε η τροπολογία. 138 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 139 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16α άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 150 και 24 ταυτόσιμες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκαν. Τροπολογία 25 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 153 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 20 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 21 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 220, άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, 200... 222. 222. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 της Επιτροπής Προϋπολογισμός. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 230. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 234. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ζήτω συγγνώμη, το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω. Αν κάποιος θέλει να αποσύρει την ψήφο του, ωραία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 242 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 248. Άρχεται η ψηφοφορία. Κοιτώ την εισηγήτρια. Λήξη της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ναι, πρέπει να είμαι προσεκτικός. 249 άρχεται η ψηφοφορία. Σε ευχαριστώ, το Όχι, συγγνώμη. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 250. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Εγώ φταίω. Εγκρίνεται. Και ναι, ναι ε, ο πρόεδρος γίνεται ρεζίλη δημοσίως. 251. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. I'll Θα είμαι πιο προσεκτικός λοιπόν. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς σε τρία-τέσσερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Το γνωρίζετε, έτσι δεν είναι. Τέσσερα πράγματα ταυτόχρονα προσπαθούσα να κάνω. Εγκρίνεται. 256. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 265 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 54 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31α άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Διακόσια εξήντα Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι, το ΕΛΚ έχει μια ψήφο παραπάνω. Ωραία, εντάξει τώρα, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 323 όχι, λάθος. Συμβαστική 37 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 3.27. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 328. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 329. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 70 ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 330 έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 331. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική 1. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 79 και 80 είναι πανομοιότυπες. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. 83. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε λοιπόν στην συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. <clears throat> Τροπολογία 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της, ψηφο... της ψηφοφορίας. Η 89 εγκρίθηκε, άρα την ψηφίσαμε την 92. Ναι, η 92 θα ψηφιζόταν μόνο σε περίπτωση που ε, εγκρινόταν η 89. Κάναμε την τροπολογία 4, ε, τη συμβιβαστική τροπολογία 4, οπότε περνάμε στην 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Συμβαστική 6. Άρχεται η, η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας Εγκρίνεται τροπολογία 108. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. 119. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 122. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. 123 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 125 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 όχι, απορρίφθηκε, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την 11, τροπολογία 11, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 130, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 13, άρχεται ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική 14, έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Είναι όμοιες οι 14 και 133 έναρξη ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνονται. Συμβαστική 15, άρχεται η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, άρχεται η ψηφοφορία, λήξη. Εγκρίνεται. 5 της Επιτροπής Προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 44 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Χόλμαϊερ. Η κυρία Χολμάγερ, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους ε, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές ε, για το πολύ επικοδομητικό κλίμα και ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τη βοήθειά της. Uh, Περνάμε στο Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Έκθεση Τάνια Φαγιών. Θέλεις το λόγο, Τάνια. Έχουμε μια, ένα αίτημα προφορικής τροπολογίας. Τον κύριο Κοέλιο. Ναι, εδώ είναι. Σύμφωνα με τον κανόνα 196. Θέλετε, κύριε Κόλλη, να διαβάσετε μόνο σα ή να διαβάσω εγώ. Πρέπει να αποφασίσουμε αν τη δεχόμαστε καταρχήν. Είναι η εξή στο άρθρο 11. Η συνεισφορά του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 85% των επιλέξιμων δαπανών ε, και το ΑΕΠ να είναι χαμηλό, της χώρας να είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου ΑΕΠ της, ε, χώρας, ε, ε Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τα άλλα θα, δεν θα ξεπερνάει το 75%. Δέχεστε αυτή την πρώτο, την, μπορούμε να δεχτούμε αυτή την τροπολογία. Καμία, καμία αντίρρηση. Θα την ψηφίσουμε πριν από την 52. Τροπολογία 36, 59 και 66 από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβασμός στο άρθρο 1. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σημαντική πρόταση στο άρθρο 3. Όχι. Ε, τροπολογία 192. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 193, στην 193. 193. 193. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική στα άρθρα 3 και 3α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Στο άρθρο 4, συμβαστική στο άρθρο 4, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 214 και 44 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 215. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 2.16. Έναρξη. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 217. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση στο άρθρο 5. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 220. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 221. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άφετ 12. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Budget 16. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Budget 17. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία επί του άρθρου, του δημοσιονομικού άρθρου 7. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 8. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί του άρθρου 9. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί του άρθρου 10. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα του κύριου Κοέλιο, όπως θα στη διάβασα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 240. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 241. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση του άρθρου 12. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για τα άρθρα 13 και 14. Έναρξη. Σελίδα 12 της δικής μου, ε, του δικού μου κειμένου. Εγκρίνεται. Τροπολογία 271. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 15. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 279. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση για το άρθρο 20. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 22. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ανθρωπολογία 287 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 23 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 24 έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 25. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 26. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 27. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 28. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 29. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 30. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράρτημα 1. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράρτημα 2. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράρτημα 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 369 και 99 που είναι ταυτόσιμες έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται, απορρίπτονται. Τροπολογία 370 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράρτημα 4, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράρτημα 5, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράρτημα 6, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράδειγμα 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το παράδειγμα 8. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας υπαριθμόν 1. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, 125, ε, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Τροπολογία ΑΦΕΤ 2, έναρξη. Έναρξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Έναρξη. Λέξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 126. Ε, Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. συμβαστική για το εκτιμώντα υπαριθμό 4. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 7 έναξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 8 και 8α νέο έναξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 9 Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 10. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για τα εκτιμώντας 11 και 12. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 15. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμάδο 17. Έναρξη. Λήξη. Συμβαστική για το εκτιμώντας 18. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 19. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 20. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 155. Ε, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 22. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 160. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία budget 4, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το εκτιμώντας 16, 26, συγγνώμη, υπέρ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Budget 5, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία για τα 34 και 34α νέο. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 164. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 165. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άφε 4. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο εκτιμώντα 33 και 34 και 34 αλφα νέο. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 170. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για, τα εκτιμώντας 37 και 38 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Budget 8 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για τα εκτιμώντα 40, 41 και 42. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 43. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 45. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 46. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 49. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντα 52. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 55, 56 και 57. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 58. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική... όχι. Budget 12. Έναρξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το εκτιμώντας 60. Λίγη ισοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο έναρξη. Ψήφισατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 41 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, 2 εποχέ. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Thank you, colleagues. Now we go straight now to... Να περάσουμε στην διελειτουργικότητα. Ah, sorry. No, we don't. We go... Όχι, δεν περνάμε εκεί. Πηγαίνουμε στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Sorry, AMIF is such a special file that it had I got it specially delivered. It wasn't in my normal. Uh, Μου το έδωσαν ξεχωριστά και δεν το είχα στο φάκελο και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Σχέδιο λοιπόν έκθεσης ε, για κανονισμό σε σχέση με τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευση. Μύρια Μτάλη, η δεν θέλει το λόγο. Πηγαίνουμε στην συμβιβαστική για την αιτιολογική αναφορά 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε Στη συμβιβαστική για τον τίτλο και την ατολική σκέψη 48 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για τα άρθρα 1 και 10 αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 2 αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο C. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίζουμε από κοινού όλες αυτές τις τροπολογίες. δηλαδή από την 297 ως την 452 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε αυτό το μπλοκ τροπολογιών. Τροπολογία 453 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και πηγαίνουμε στην συμβιβαστική για το άρθρο 3 και τις ατολικές σκέψεις 12, 13, 14 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Και πηγαίνουμε στη συμβιβαστική για το άρθρο 3α νέο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 4. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Τροπολογία 52 πηγαίνουμε. Στην σελίδα 8 της δικής μου λίστας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 52. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα συμβιβασμός για το άρθρο 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στο άρθρο 6 παράγραφο 3 και στην τροπολογία 3, 4, 9. 3.50 και 56. Δηλαδή 3.49, 3.50 και 56 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνονται. Πηγαίνουμε στην 352, όχι δεν πηγαίνουμε εκεί, πηγαίνουμε στη συμβιβαστική για το άρθρο 7, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πηγαίνουμε στο συμβιβασμό για το άρθρο 8, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη συμβιβαστική για το 51α, το άρθρο 9, χωρίς την παράγραφο 2 και χωρίς την παράγραφο 6, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 9, παράγραφος 2, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστή για το άρθρο 9 παράγραφο 2 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτε, απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα στη συμβαστική για το άρθρο 9 παράγραφος 6 και αιτιολογική σκέψη 17 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στο άρθρο 11, παράγραφο 1, σημείο A. Τροπολογία 391 και 392. Ναι. ...391-392 από κοινού ψηφίζουν. Πέρασε. Απορρίπτονται. Συμφιβασμός για το άρθρο 12 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα, συγκρίνεται. Συμβιβαστική στο άρθρο 13 χωρίς την παράγραφο 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Συμβιβαστική στο άρθρο 13 παράγραφος 1 τμήμα 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική το άρθρο 13 παράγραφος 1 τμήμα 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. μεβαστική για το άρθρο 14 και τη Συντολική Σκέψη σκέψεις 34-35. Άρχεται η ψηφοφορία. Να σηκώνει και λίγο πιο ψηλά για να καταλαβαίνουμε, Μύρια, αν είναι υπέρ ή κατά αυτό που λες. Ωραία, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη συμβαστική το άρθρο 15 και την εντολική σκέψη 31. Άρχεται η ψηφοφορία. And the Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 16 και την ατολική 11α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 17 και η τολική σκέψη 38 ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική το άρθρο 17α νέο άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική το άρθρο 18 και το 40 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική τώρα το 20 και, το, και την σκέψη 41 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική για το άρθρο 21 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική για το άρθρο 25 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 26 και το σκέψη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 467. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 από, από την Επιτροπή Προπολογισμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 468. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 29. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 30 και την ετολική σκέψη 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 490. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Σε για το 32 και τη σκέψη 56 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το παράρτημα 1 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 528 άρχεται ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το παράρτημα 2 και τελικές σκέψεις 7, 8 και 9. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το παράρτημα 3 και την ετολική σκέψη 5β ναι, Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το παράρτημα 3, σημείο 4α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται Η τροπολογία 660 και 661 είναι ταυτόσιμες. Από κοινού τις ψηφίζουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβιβαστή για το παράρτημα 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται συμβιβαστική για το παράρτημα 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 683. 684 μάλλον. Πέρας. Συμβιβαστική για το παράρτημα 8 άρχεται ψηφοφορία περασε Εγκρίνεται. 165 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 164 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 166 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σερευαστική για την εντολική σκέψη 2. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 169. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 170. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 171. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για την Ανατολική Σκέψη 4, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 100 όχι. Ντεβε 2, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, γκρίνεται. Ντεβε 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για την εντολική σκέψη 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Κοντεύουμε. Εγκρίνεται συμβαστική για την 5α νέα αιτιολογική. Πέρασε. Εγκρίνεται. 178. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒ 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική για την αιτιολογική σκέψη 18 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 19 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 220 άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 13 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 221 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 222 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 223 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4 της Επιτροπής Προπολογισμού άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, όλοι είμαστε κουρασμένοι. Δεν την ψηφίζουμε την budget 4, όμως να κυρώνω αυτή την αλλά δεν το πρόσεξε και κανεί. Έτσι που είναι όλοι κουρασμένοι. Λοιπόν, συμβιβαστική για τι αιτιολογικέ σκέψει 21-22 άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Εγκρίνεται. Κοντεύουμε 2.30. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλο πάντων, υποτίθεται ότι κοντεύουμε, έτσι το λέω. Για να μην χάσετε το ηθικό σας. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 232 τροπολογία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το 24, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 238-239 ταυτόσιμες, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. ΔΕΒΕ 17 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 18 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 241, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 243, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο 27α νέο, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο 27β νέο, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 249-250. Απορρίπτονται. Τροπολογία 26, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.51, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο αιτιολογικό 30, άρχεται. Η ψηφοφορία πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική συντολογική 32 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική συντολογική 33 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στην αιτιολογική 37 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε εγκρινεται τροπολογης Τροπολογίες 34-277. ταυτός μεσάρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 278 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 279 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 283. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 284. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. ΔΕΒ 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική για το Recital 55, άκτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και συμβαστική για το Recital 58, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ, 23 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έχουμε δύο ακόμη σύντομες, σύντομες ψηφοφορίες. Παρακαλώ. Παραμείνετε. Κοντεύουμε. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγητής ο κ. Μέλο. Θέλετε το λόγο. Ε, έχω τυφλωθεί που βρίσκεστε. I'm, I'm really sorry. I think it's it should be uh, Jerome first. No, no, but I think there's a protocol kind of order. Υπάρχει πρωτόκολλο εδώ, ε, εθιμοτυπία. Πρέπει να είναι πρώτος, να πάει πρώτος ο Γερόν. Ξεκινάμε με τη διαλειτουργικότητα, σύνορα και θεωρήσεις. Συζητητής ο Γερόν Λέναρς. Θέλεις το λόγο, όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόκειται για το κείμενο στο οποίο συμφωνήθηκε για τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων ονομαστική ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, 43 ε, ψήφοι υπέρ, 11 κατά, 0 απόχέ. Συγχαρητήρια κύριε Λέναρ. Και θα ψηφίσουμε τώρα το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, κύριος Μέλος, ηγητή, θέλετε το λόγο. Όχι, ωραία. Περνάμε κατευθείαν λοιπόν στην ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ονομαστική. The vote is uh, closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, καμία αποχή. Σα συγχαρητήρια κύριε Μέλο. Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε στις 4 και 4. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.